συνάδελφοι, θέλω να σας καλωσορίσω στην ε, απογευματινή συνεδρία της Επιτροπής μας και χωρίς άλλη καθυστέρηση να παρουσιάσω τον ομιλητή μας, κύριο Ντάνιελ Φίωτ, από το Institute for Security Studies της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα παρουσιάσει την έρευνα σχετικά με τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας από το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η Επιτροπή μας είχε ζητήσει τη σύνταξη αυτής της έρευνας το 2018 και είχε παραδοθεί λίγο πριν τη λήξη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περίοδου. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που μπορεί να ασκήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, είναι αρκετά περιορισμένος. Περισσότερες αρμοδιότητες θα έχουν τα εθνικά κοινοβούλια, το εύρος τους όμως διαφέρει ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο του κάθε κράτους μέλους. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, το γεγονό ότι πολλά κοινοβούλια με διαφορετικό καθεστώ στο καθένα ελέγχει αυτό το νέο ταμείο είναι αρκετά περίπλοκο. Για τον λόγο αυτό θα ακούσουμε με ενδιαφέρον τις απόψει, τις δεξαμενή σκέψεις του κ. Φίωτ για τα θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλάπω. Είναι η δεύτερη φορά για τη δεύτερη μελέτη κατά σειράν. Με μεγάλη χαρά λοιπόν βρίσκομαι εδώ μαζί σας και σας ευχαριστώ για τα καλά σας ε, λόγια. Θα σας ε, δώσω μια σύνοψη της ε, μελέτης, της έκθεσης και κάποιες από τις συστάσεις ή τέλος πάντων την βασικότερη κατεύθυνση σχετικά με το EDF, EDF με και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία της μελέτης που σημειώθηκαν και σωστά. Υπάρχει το ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή ο ρόλος του Κοινοβουλίου στον έλεγχο του Ταμείου και το εθνικό επίπεδο. Στη μελέτη προσπάθησα να αφιερώσω αρκετό χώρο και στα δύο αυτά στοιχεία, σκεπτόμενος και κάποιες ε, εθνικές ε, συζητήσεις στα κοινοβούλια ως προς το Ταμείο, αλλά και ως προς την ανάπτυξη του δυναμικού, του αμυντικού και το πώς θα μπορούσε να σχετίζεται το Ταμείο αυτό με άλλες πρωτοβουλίες αμυντικές, όπως μόνιμες δομές συνεργασίας. Αυτά ως προς την αρχιεκτονική, τη δομή της μελέτης. Οι παράμετροι το πλαίσιο δηλαδή εντός του οποίου εργαστήκαμε, ε, στην εισαγωγή υπάρχει ήδη ένας περιορισμός. Δηλαδή, υπό την νομοθετική ε, ενωσιακή έννοια, εγώ εργαζόμουν επί μιας πρότασης κανονισμού για το Ταμείο. Επομένως υπάρχει ένα πλαίσιο για την συζήτηση η οποία διεξήχθη εδώ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες έννοιες, κάποιες σκέψεις που δεν είναι καινούργιε, αλλά τις βλέπουμε στην ε, βιβλιογραφία της ευρύτερη συζήτηση ε, ε, του κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα θέματα μήνυ υπό τι συνθήκε. γενικώ μιλώντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έναν σχετικά περιορισμένο ρόλο στα θέματα ασφαλείας και αμήνης. Αυτό το πρόσεξαν οι ακαδημαϊκοί μελετητές υπό δύο πτυχές. Καταρχάς, την τυχή της ε, δημοκρατικής νομιμότητος και το επίπεδο της φιλοδοξίας που έχουμε στο έργο, στο πείραμα αυτό. Έχουμε κάποιους περιορισμούς λοιπόν διακυβερνητικής προσέγγισης ως προς την αμυντική ολοκλήρωση. Πολλές μελέτες εστιάζονται στο πώς, τι ρόλο μάλλον θα μπορούσαν να διαματήσουν τα εθνικά κοινοβούλια λιγότερη εστίαση έχουν αφιερώσει οι μελετητές λόγω των χρονικών περιορισμών στο ίδιο το ταμείο, το EDF, αλλά νομίζω ότι πρέπει να χαιρετήσει κανείς την Επιτροπή που ζήτησε τη μελέτη αυτή, ώστε να δούμε τι δυνατότητες θα μπορούσαμε να έχουμε με την εισαγωγή του ταμείου αυτού. Στη δική μου έκθεση λοιπόν πολύ προσεκτικά λέω ότι οι πρωτοβουλίες όπως η PESCO, CARD και άλλα σχέδια μένουν σε μια ευρύτερα διακυβερνητική δομή. Το EDF είναι διαφορετικό δημιούργημα. Όχι μόνο γιατί χρηματοδοτείται απευθεία από τον ενωσιακό προπολογισμό, αλλά και επειδή το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη στον κανονισμό. Και επομένω υπάρχει μια συζήτηση που πρέπει να γίνει για το ποιο θα πρέπει να είναι ο κοινοβουλευτικό έλεγχο και με τι θα πρέπει να μοιάζει. Μία πτυχή τη έκθεση που είναι κάπω προβληματική και ίσω ευαίσθητη και ένα από του λόγου για του οποίου πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι ο συσχετισμό μεταξύ αφενό του Ταμείου και αφεντέρου με την μόνιμη δομή συνεργασίας. Η μελέτη μου εστιάζεται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Ταμείου, αλλά υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση για τις σχέσεις της διακυβερνητικής δομής στα θέματα αμήνης και στις πιο υπερεθνικές δομές στα ίδια θέματα και σε αυτό θα επανέλθουμε. Θα ξεκινούσα με την οπτική γωνία των Εθνικών Κοινοβουλίων και ένα από τα βασικά συμπεράσματα προκύπτει από τη μελέτη και δεν είναι έκπληξη φαντάζομαι είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα ως προς τα συμφέροντά τους στα θέματα μήνης και στα θέματα του αμυντικού ταμείου αλλά και ως προς το εθνικό επίπεδο, δηλαδή τι εμπειρογνωμοσύνη χρειάζεται ή μάλλον διατίθεται για να μπορεί να ελέγχονται οι πρωτοβουλίες αυτές. Αν κανείς έχει αντίγραφο της μελέτης θα δει ότι η απόπειρα του να δει, εξετάσει τις συζητήσεις τις κοινοβουλευτικές που διεξιάγονται και αυτή η μελέτη ε, πολύ σωστά ο πρόεδρος είχε πει ότι δημοσιεύθηκε πριν από λίγους μήνες και ίσως δεν αποτυπώνει λοιπόν τις αλλαγές ε, που έχουν λάβει χώρα από τότε μία από τις πιο σημαντικές παρατηρήσεις υπό την έννοια των εθνικών κοινοβουλίων είναι όχι μόνο η ασύμετρη πληροφορία μεταξύ της συζήτησης που διεξάγεται στις Βρυξέλλες και στο εθνικό επίπεδο. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις υπήρχε ιδιαίτερα σημαντική έλλειψη πληροφορίας για τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά επίσης ανάλογα με το ποιο είναι το Εθνικό Κοινοβούλιο για το οποίο συζητούμε, υπήρχε σε κάποιο βαθμό μια δυσκολία κατανόησης του πώς το EDF από, κοινού με την ΠΕΣΚΟ και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες θα επηρεάζει τις εθνικές πρωτοβουλίες στις αμυντικές δαπάνες. Και για τον εξοπλισμό που θα μπορούσε να ενδιαφέρει την συγκεκριμένη χώρα, για παράδειγμα. Ένα από τα στοιχεία λοιπόν που ανακύπτουν από τι συζητήσει στι Εθνικές και μπορεί να ισχύει και για την ευρύτερη συζήτηση είναι η σχέση ή μάλλον ο ορισμός του τι ακριβώς σημαίνει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε διότι αυτό που είναι σαφές από την ανάλυση στα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ότι διεξάγονται κάποιες συζητήσεις εκεί που εστιάζονται περισσότερο στην παρακολούθηση της πολιτικής, δηλαδή υπήρξε μια δικασία κοινοβουλευτικών επιτροπών να συλλέξουν τις περισσότερες πληροφορίες που μπορούσαν από τα αρμόδια υπουργεία, από γραμματείες, από εμπειρογνώμονες. Παρακολούθηση λοιπόν, επιτήρηση. Κάποια κοινοβούλια πήγαν και πέραν αυτού, δηλαδή τον έλεγχο παρακολούθησης, πήγαν περισσότερο σε εκείνο που θα αποκαλούσε κανείς ή το κάνουν οι ακαδημαϊκοί πολιτικός έλεγχος. Δηλαδή τι δυναμικό πρέπει να αναπτυχθεί ενωσιακά. Πώς θα πρέπει να συνεισφέρει το EDF στη συνδιαμόρφωση της αγοράς της αμυντικής. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες προτεραιοποίησης αυτού του δυναμικού σε εθνικό επίπεδο. Στις αναλύσεις λοιπόν των Εθνικών Κοινοβουλίων υπάρχουν μόνο δύο είδη διαλόγου συζήτησης. Ας συλλέξουμε πληροφορίες αφενός και αφετέρου ας σκεφτούμε πιο στρατηγικά. EDF, PESCO και άλλες πρωτοβουλίες πώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εθνική συζήτηση για την ανάπτυξη του δυναμικού για τις προμήθειες τα αμυντικές. Πηγαίνοντας περισσότερο στο ενωσιακό επίπεδο και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είπα από την αρχή, υπήρξε ένας κάποιος περιορισμός σχετικά με τις πηγές που είχα στη διάθεσή μου. Εγώ εργαζόμουν στα πλαίσια της πρώτης κανονισμού. Και εκεί έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε για το, την περιοχή στην οποία θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό έλεγχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαβάζοντας την πρόταση ως έχει σήμερα προκύπτει με σαφήνεια ότι το Κοινοβούλιο τουλάχιστον θεωρητικά έχει μεγάλο δυναμικό συμμετοχής στον έλεγχο του Ταμείου πέραν της εμπειρίας που υπάρχει σε παραδοσιακά πλαίσια CSDP που είναι περισσότερο διακυβερνητική η προσέγγιση είναι συνομοθέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιλούμε προφανώς για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και εν ώψη των συζητήσεων ΠΔΠ και το Κοινοβούλιο έχει ρόλο εδώ να διαματίσει. Το ζήτημα είναι ποιος πρέπει να είναι αυτός ο ρόλος και πού πρέπει να εστιάζεται, αν πρέπει. Διαβάζοντας λοιπόν την πρόταση στενά, κατά γράμμα, υπάρχουν δύο δυνητικές περιοχές που μπορεί να υπάρξει αυτή η επιτήρηση, αυτός ο έλεγχος. Στο τέλος του επταετού κύκλου λειτουργίας, κατά πόσο δηλαδή το Ταμείο έχει επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την στρατηγική αυτονομία κτλ. Και οι ετήσιες αξιολογήσεις, εκτιμήσεις του κατά πόσο το Ταμείο επιτυγχάνει τους τρέχοντες στόχους του. Επομένως έχουμε δύο χρονικές φάσεις. Ένας επταετής κύκλος και ένας ετήσιος. Αυτό που δεν είναι απολύτως σαφές από αυτό το πλαίσιο των πραγμάτων και δεν θα μπορούσε να το επεξεργαστεί κανείς περαιτέρω στη μελέτη είναι πώς αυτό πρέπει να εκφράζεται. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να συμμετέχει χρονικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετησίως και πώς στο τέλο στο τέλος του επταετούς κύκλου. Και το πρώτο ερώτημα που προκύπτει νομίζω στα συμπεράσματα με σαφήνεια είναι μια έκκληση, πρόσκληση, όχι να σκεφτούμε απλώς Ποιε θα πρέπει να είναι οι αρμοδιότητες ελέγχου του Κοινοβουλίου, αλλά και με ποια στόχευση για ποιους σκοπούς. Ίσως να ακούγεται προκλητική αυτή η ερώτηση, αλλά είναι επίτηδες που έχει διατυπωθεί έτσι. Δηλαδή πρέπει απλώς το Κοινοβούλιο να προχωρεί σε μια εκτίμηση του κατά πόσον το Ταμείο πράγματι επιτυγχάνει τους βασικούς του στόχους ή θέλουμε πολύ πιο ουσιαστική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ορισμό του δυναμικού, στα προγράμματα εργασίας. Αυτή η ερώτηση είναι ανοιχτή και πρέπει να ασχοληθούν με, αυτή, και τα μέλη, οι βουλευτές. Τι σημαίνει λοιπόν κοινοβουλευτικός έλεγχος. Οποιαδήποτε απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι εξορισμού πολιτικά ευαίσθητη και σχετίζεται με το πώς βλέπει τον εαυτό του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη δυναμικού προς το μέλλον, για μελλοντικές τεχνολογικές τάσεις. Ένα από τα σημεία που αναφέρω στην έκθεση είναι η στάση του Κοινοβουλίου σε σχέση με μελλοντικές τάσεις της τεχνολογίας. Αν θέλουμε δηλαδή να επενδύσουμε το 5% σε τεχνολογίες εχμής, έχει μια σαφή τοποθέτηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούμε ως προς αυτές τις τεχνολογίες. Υπάρχει ηθική διάσταση ως προς αυτές. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει και το Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια. και δεν είναι σαφές σε κάθε περίπτωση ότι οι συζητήσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια εισέρχονται σε τόσο ουσιαστικά οι ευαίσθητα θέματα για το πώς ορίζει κανείς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ποιο, ποια είναι η απόλυξη αυτής της διαδικασίας ελέγχου. Άλλο ένα στοιχείο που εξετάζω στην έκθεση και δεν είναι καθόλου εύκολο προς ανάλυση ή προς συζήτηση είναι η σχέση μεταξύ αφενός του EDF και αφετέρου της ΠΕΣΚΟ. Ή για να το πούμε πιο ακαδημαϊκά ή ερευνητικά, ποια είναι η σχέση μεταξύ μιας υπερεθνικής προσέγγισης και μιας διακυβερνητικής προσέγγισης. Τεχνικώς μιλώντας, θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί και ποια είναι η σχέση μεταξύ του EDF και της μόνιμης δομής συνεργασίας πώς σχετίζονται, πώς συνεργάζονται, πώς θα έπρεπε να διεξάγεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος εκεί. Επίσης, Ένα ερώτημα είναι και ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή θα προχωρήσει προς την προτεραιοποίηση για τα θέματα αυτά. Έχει πει η Επιτροπή ότι θα λάβει υπόψη της τα συμπεράσματα του σχέδιου ανάπτυξης δυναμικού και εντός δυναμής αυτής η Επιτροπή θα έχει μια άμεση επικοινωνία, ανοιχτή γραμμή με τα κράτη-μέλη για τα χαρτοφυλάκια που θα ορίζονται υπό το EDF. Επομένως, μιλώντας για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, μιλούμε επίσης για την ασυμμετρία της πληροφορίας, τι πληροφορία έχει κανείς σε πολύ τεχνικά ζητήματα, όπως οι αμυντικές προμήθειες και η ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και πώς σχετίζονται όλα αυτά μεταξύ διακυβερνητικής ολοκλήρωσης και υπερεθνικής. Το Κοινοβούλιο λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τα εξετάσει όλα αυτά. Για να μην μακρηγορήσω, ίσως θα μπορούσα να πάω τώρα σε κάποιες από τις συστάσεις και εδώ όταν συνέτασα την έκθεση αυτή το διαθέσιμο υλικό για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο κανονισμός, ποια θα ήταν η δομή, ήταν πιο περιορισμένο το πλαίσιο αυτό από ό,τι είναι σήμερα. Αλλά πιστεύω ότι κάποιες από τις συστάσεις μου δίνουν τροφή προσκέψη. Αυτή η συμμετρία της πληροφορίας που ανέφερα. Δεν πρέπει να υποτιμά κανείς το επίπεδο της εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για να ελέγξει αποτελεσματικά κανείς την καινοτομία στην αμυντική έρευνα. Ίσως να γνωρίζετε κάποιοι από εσά ότι ακόμα και εντός του οργανισμού αμήνης μία από τις πιο σημαντικές πτυχές ώστε να έχει κανείς εσωτερικά την εμπειρογνωμοσύνη για να χειρίζεται, να διαχειρίζεται υψηλά τεχνικά έργα και αυτό σίγουρα θα κατευθύνει τις κατευθύνσεις για τη δημιουργία μιας νέας γάμα δέλτα ε, που θα καλύπτει αυτά τα θέματα. Αυτές οι πτυχές δεν πρέπει να χαθούν από την εξέταση, την ανάλυση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εκεί κάνουμε και μία σημείωση για το ρόλο της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ. Εάν θέλετε, επιθυμείτε να έχετε αποτελεσματικό έλεγχο και να τον ενισχύσετε για τα θέματα αμήνης, θα πρέπει να δείτε τη βάση εμπειρογνωμοσύνης που έχει στη διάθεσή σας για να τα διαχειρίζεστε όλα αυτά. Και δεν μιλάω μόνο για τους βουλευτές, για τα μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες, οι οποίες είναι αποτελεσματική σημασίας για να ορίζει κανείς τις προτεραιότητες και το δυναμικό αμήνης. Η δυνατότητα λοιπόν πληροφορίας, συλλογής πληροφορίας και διαχείρισής της είναι πολύ σημαντική και αυτό οδηγεί και στο καθεστώς της COSAC και της IPC. Οι σχέσεις μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και η σχέση με το CFSP. Και για να το πω αυτό διακριτικά και λεπτά, το δυναμικό και των δύο αυτών φορέων δομών δεν, έχει, δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί πλήρως. Θα το πω έτσι. Εξέτασα κάποιες από τις ανταλλαγές απόψεων που έχουν λάβει χώρα στα δύο αυτά σώματα και ίσως μπορεί να μπει κανείς ότι είναι κάπως επιφανειακές. Οι συζητήσεις αυτές είναι ένας τρόπος networking, διαδικτύωσης μεταξύ κοινοβουλευτικών επιτροπών, οπωσδήποτε, αλλά πώς μπορεί κανείς να πάει πιο πέρα η απλή ενημέρωση των βουλευτών για το ποιο είναι το θέμα της συζήτησης σε μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τις τεχνικές διαστάσεις και την πολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ κρατών μελών είναι απόλυτα σημαντική. Ε, ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα κράτη-μέλη. Κόσακ λοιπόν και IPC, πώς αυτά μπορούν να γίνουν στρατηγικά πιο σημαντικά ώστε να αυξηθεί και πάλι η δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου και για τις ε, ε, τεχνολογίες αυτές εχμής και τις μελλοντικέ τάσεις. Και αυτό βεβαίως είναι μια πολύ λεπτή συζήτηση. Όλοι γνωρίζουμε την συζήτηση για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα, αλλά η δυνατότητα άσκηση ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων εξαρτάται από το βαθμό της, του προσανατολισμού, της κατεύθυνση αυτής της συζήτησης, όχι μόνο από την έννοια των επενδύσεων, αλλά και γιατί. Γιατί να επενδύσουμε σε αυτές τις τεχνολογίες. Με ποιο στόχο. Ε, θα έμενα εδώ. Νομίζω ότι έχω δώσει αρκετά στοιχεία για μια Καλή συζήτηση και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φιώτ. Ε, και έχουμε τώρα κάποιες ερωτήσεις. Το λόγο έχει πρώτο ο κύριος Ριβιέρα. Euh, euh. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την ε, παρουσίαση. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται την πρόκληση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ε, πραγματικά επιβεβαιώνει την άποψή μου ότι ε, με αυτό το ταμείο και τη δημιουργία αυτού του ταμείου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπέρασε τα όρια διότι αυτά δεν είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών της Ένωσης και επίση έχασε και την κοινή λογική. Ε, η Κομισιόν χρηματοδοτεί αναζήτηση προγραμμάτων σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και ε, ε, έτοιμα προς τους, ε, τις ένοπλες δυνάμεις. Στη Γαλλία είχαμε, για παράδειγμα, ε, Συμβάσει ε, με το στρατιωτικό σκέλο. αν δεν υπάρχει κάποια στρατηγική απάντηση ενός ευρωπαϊκού στρατού, ε, όταν δεν υπάρχει ευρωπαϊκό στρατός και δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό στρατός, είναι σαν να χάνουμε την αίσθηση της κοινή λογικής και ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία αποτελούν ένα στόχο να προωθήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι όλο ένα και πιο φεντεραλιστικό. Ε, νομίζω ότι αναφερθήκατε και στα εθνικά κοινοβούλια και είπατε ότι υπάρχει ένα όρομα της άμυνας που είναι τελείως διαφορετικό και νομίζω ότι αυτό βολεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θα επιτρέψει ε, ε, στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια να μπορέσουν να έχουν τελικά μία ενοποιημένη ε, άποψη ε, για το τι ακριβώς ε, ζητούν τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι το οποίο δεν αναφέρεται και δεν είχατε χρόνο ίσως να ε, αναφέρετε είναι τι γίνεται με τη χρήση αυτών των κονδυλίων του Ταμείου. Υπάρχουν δύο στοιχεία. Αυτό το οποίο είναι λυπηρό είναι ότι τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να περάσουν από μια συνεργασία τουλάχιστον τριών κρατών, ενώ σε πολλά άλλα προγράμματα διμερού συνεργασίας ε, είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία και μας επέτρεψαν να έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Πώς μπορούμε τώρα να επιβάλλουμε τρεις χώρες οπωσδήποτε. Ε, γιατί όχι δύο χώρες που συνεργάζονται ε, να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Θα πρέπει να βρουν κάποιον τρίτο ε, για να κάνουν συνεργασία. Αυτό σημαίνει ότι σπαταλούμε πόρους τελικά. Και επίσης ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια και από ξένες δυνάμεις. Ε, ξέρω ότι ε, οι άμεσες θηγατρικές επιχειρήσεων δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια ακόμα και αν έχουν θηγατρικές στην Ευρώπη, αλλά επιχειρήσεις οι οποίες είναι ε, εγκατεστημένες στην Ευρώπη από το 1994, αν δεν κάνω λάθος, θα μπορούν κάλλιστα να ε, χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια και θα μπορούν να το κάνουν και χώρες, επιχειρήσεις οι οποίες είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματοδοτούμε δηλαδή έρευνα και ανάπτυξη η δεν είναι προ το συμφέρον αυτού που πληρώνει ε, για την έρευνα και την ανάπτυξη αυτή στην άμυνα, δηλαδή του Ευρωπαίου πολίτη. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που ήρθα κάπως καθυστερημένος ε, στην παρουσίαση, αλλά διάβασα και το έγγραφο για την έκθεσή σας και πρόσεξα και αυτό που είπατε στο τέλος για το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εγώ έχω κάποιες επικρίσεις διαφορετικής φύσεως ε, ε, από τις επικρίσεις ε, του συναδέλφου με τις οποίες δεν συμφωνώ απολύτως παρεπιπτόντως. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό να λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί πράγματα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αντιθέτως για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι γνωρίζει, ότι ξέρει ότι μπαίνει σε χωράφια τα οποία της είναι κάπως άγνωστα και δέχτηκε την εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών και της βιομηχανίας. Και το μοντέλο το οποίο έχει ε, συσταθεί προς το παρόν για τη χρήση αυτών των κονδυλίων είναι ένα πάρα πολύ καλό μοντέλο, στο οποίο προς το παρόν θα πρέπει βέβαια να επαγρυπνούμε, αλλά ε, φαίνεται να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Και η βιομηχανία φαίνεται να είναι ικανοποιημένη αρκετά, τα κράτη-μέλη προς το παρόν είναι αρκετά ικανοποιημένοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τη δουλειά δουλειά της χωρίς να ε, στερηθεί και δυνατότητα νέων πρωτοβουλειών. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι το μοντέλο αυτό δεν λειτουργεί και πολύ άσχημα, αρκετά καλά λειτουργεί. Θα πρέπει να δούμε βέβαια και τι γίνεται με τη γραφειοκρατία, με τον αυτόματο χαρακτήρα ε, των ε, θεμάτων των οποίων, τα οποία απασχολούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα. Και ε, εδώ είναι και κάτι σημαντικό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω. Το Ταμείο για την Άμυνα είναι μια πρόοδος από πλευράς αρχών αλλά δεν αλλάζει και τα πράγματα ε, εκ βάθρων. Δεν είναι ε, game changer που λέμε στα αγγλικά. Είναι σταγόνα στον ωκεανό το προπολογισμό που προσφέρεται σε σχέση με τον προπολογισμό που σκοτωδεύουν ε, για την άμυνα οι χώρε μέλη. 13 δι σε 7 χρόνια. Ε, ο προπολογισμό άμυνας τη Γαλλία είναι 34 δι ευρώ. Ε, Επομένως, ε, αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, ε, το οποίο είναι και συνεργατικό αν θέλετε, ε, έχει και ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι εμβρυϊκό σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος. Υπάρχουν κάποιοι που επικρίνουν και λένε προσέξτε ότι είναι κάτι το οποίο θα ξεφύγει τελείως από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Κάποια στιγμή πρέπει να μην προσπαθούμε να υπερβαίνει η αρχή του κοινοβουλευτικού ελέγχου ε, από τα όσα έχει να προσφέρει αυτό το ταπεινό πρόγραμμα. Είναι σαν να μην, βάζουμε, να μην ιεραρχούμε σωστά τις προτεραιότητές μας. Ε, ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να μην είναι ο βέλτιστος δυνατός ή στα πρότυπα που θα ήθελαν κάποιοι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, σκέφτομαι ε, τις εκτελεστικές και τις κατεξουσιοδότηση πράξη. Αυτά είναι τεχνικά θέματα όμως. Ε, είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά ε, ε ταπεινή ως προσπάθεια ε, οι χώρες μέλη και οι βιομηχανίες ε, θα απομακρυνθούν από το Ταμείο αν το Ταμείο δεν είναι εύκολο στη χρήση του. Και αν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ε, διαπιστώσουν ότι πρόκειται για μια γιγάντια γραφειοκρατία στην οποία ο κοινοβουλευτικό έλεγχος είναι υπερβολικό σε σχέση με τις πραγματικές προκλήσεις, τότε θα αποδεσμευθούν και θα κλείσουν την πόρτα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνα και ο κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν θα έχει κανένα νόημα. Πρέπει λοιπόν να ιεραρχήσουμε σωστά τι προτεραιότητέ μα. Και εδώ ολοκληρώσω και με δύο πολύ μικρές παρατηρήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε μου, και ε, μάλιστα είναι και φημισμό ε, να επισημαίνετε δύο πράγματα. Πρώτον, η έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διεκδικήσει ε, απόλυτο κοινοβουλευτικό έλεγχο για αυτή την πρωτοβουλία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μπορεί να, να αποδείξει ότι όντως ε, μπορεί να μιλήσει για κάποια θέματα άμυνας. Ε, είμαι και εγώ ένοχο ε, και εγώ ε, προέδρευα και σε αυτή την υποεπιτροπή. Δεν αποδείξαμε ότι έχουμε την αξιοπιστία και την εμπειρογνωμοσύνη μέχρι τώρα συλλογικά ως σώμα. Δεν είμαστε ένα όργανο το οποίο μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και υπάρχουν καλοί λόγοι γι' αυτό, για ε, το λόγο για τον οποίο δεν μας λαμβάνουν υπόψη οι σοβαροί παράγοντες της αγοράς της άμυνας. Ε, δεν έχουμε εμπειρογνωμοσύνη, μπορεί να την αποκτήσουμε, προς το παρόν όμως μας μένει αρκετή δουλειά. Και για το πεδίο τη αρμοδιότητάς μας. Γιατί εδώ σε αυτή την υποεπιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας αρέσει να ασχολούμαστε και να έχουμε άποψη επί παντού επιστητού, αλλά σε ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε να έχουμε αρμοδιότητα και εμπειρογνωμοσύνη ε, και ε, απέναντι στα εθνικά κοινοβούλια, ε, κυρίως για αποστολές ε, ασφάλειας και άμυνας, ε, πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ακόμα ότι έχουμε την εμπειρογνωμοσύνη. Για παράδειγμα, γίνονται κάποιες επιχειρήσεις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα πόρα απέχουμε από κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δούμε βέβαια και τι γίνεται με τη διακοινοβουλευτική διάσκεψη και την ΚΟΖΑΚ. ακόμα είναι... Αυτά τα πράγματα πάρα πολύ περιορισμένα. Εγώ συμμετείχα στη συζήτηση πολλές φορές. Δεν έχω δει καμία επιχειρησιακή συζήτηση ε, που θα δείχνει ότι υπάρχει ουσιαστική δουλειά και συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Κάποιες φορές ε, συζητάμε κάποιες ε, ε ωραίες συζητήσεις, πνευματικό επίπεδο κλπ. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι επιχειρησιακό ε, κοινοβουλευτικό έργο για κάτι το οποίο θα έπρεπε εγώ να ελέγχω περισσότερο. Τώρα, η άμυνα, αν είναι στρατιωτική, αν είναι ο, κλάδος, η βιομηχανία, αν υπάρχει υπουργό άμυνας ενός κράτου μέλους, αν παρακολουθήσει τις, εργασίες της ε, ε, συνέλευση θα φύγει κλαίγοντα. Ε, πραγματικά θα συνεχίσουν να συζητάνε σοβαρά όλα αυτά τα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν του δίνουμε καμία εξουσία. Ε, Επομένω, το μπαλάκι είναι και στο γήπεδό μα. Ε, αν θέλουμε να έχουμε περισσότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο και να φωνάζουμε ότι πρέπει να έχουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε και την εμπειρογνώμοσύνη και την αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Sorry, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Δεν άκουσα το όνομά μου. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της μελέτης. Νομίζω ότι ο κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι ένα σημαντικό τμήμα, από τα πιο σημαντικά τμήματα τη εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, έχουμε τι κατεξοδότησε πράξει και το Κοινοβούλιο έχει τρει μήνε για να αξιολογήσει ένα σχέδιο προγράμματος και να το σταματήσει. Αλλά δεν ενεκρίθη αυτός ο, η δυνατότητα ελέγχου, ο μηχανισμός ελέγχου, όταν ολοκληρώνονταν οι διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Άμυνας. Η Επιτροπή που είναι αρμόδια, η Ήτρε, μετά τις εκλογές όμως επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι η πρόθεσή μας. Τι άλλες δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου θα είχαμε, γιατί ξέρουμε ότι 13 δις είναι η χρηματοδότηση, άρα πρέπει κάπως να ελεγχθεί η χρήση των πόρων αυτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Φίωτ, για αυτά που είπατε. Όντω, τη διάβασα τη μελέτη σα και παρακολούθησα με ενδιαφέρον αυτά που μα είπατε. Θα είχα διάφορε ερωτήσει να σα κάνω. Αλλά, καταρχά, αυτό που είναι ενδιαφέρον, λέτε στη μελέτη σας, ότι φαίνεται σαν να μην έχει κανένα σαφή ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη λειτουργία του Ταμείου Άμυνας και ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν είναι σε θέση να παίξουν το ρόλο τους σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουν σαφείς αρμοδιότητες γι' αυτό. Επίσης διαπιστώνεται ότι παρόλα αυτά τα κράτη-μέλη έχουν δικαίωμα βέτο, de facto. Οπότε τίθεται το ερώτημα. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ένα, τη δυνατότητα πολιτικού ελέγχου της λειτουργίας του Ταμείου Άμυνας και με κάθε σεβασμό θέλω να σας πω ότι αυτό που μας λέτε ότι δεν έχουμε αρκετή εμπειρογνωμοσύνη δεν, δεν αρκεί ως δικαιολογία. Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα πολιτικό θέμα. Υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση. Αυτό κάνει η πολιτική. Πρέπει να ελέγχει κατά τη γνώμη μου τέτοια θέματα. Δηλαδή τη λειτουργία τέτοιων οργανισμών και τη χρηματοδότηση. Όμως περιορίζεται η δυνατότητά μας μόνο στο καθορισμό της χρηματοδότησης μέσω του, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και μετά τελειώνουμε. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα. Αυτό λέτε. Αυτό πραγματικά λέτε πάνω κάτω. Δεύτερον, στη Γερμανία. Για τα μεγάλα προγράμματα, εάν για παράδειγμα η πρικοδότηση είναι πάνω από 25 εκατομμύρια, τότε υποχρεωτικά η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πρέπει να συμμετάσχει στη λήψη της απόφασης. Δεν θα ήταν αυτό μια δυνατότητα. Να κάνουμε κάτι παρόμοιο για τα σημαντικότερα προγράμματα. Πώς το αντιμετωπίζετε θα ήταν πολύ καλό πιστεύω να κοιτάξουμε το γερμανικό μοντέλο να δούμε αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και τρίτον, στη μελέτη σας διάβασα ότι διαπιστώνετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει μεγάλο ρόλο, τα εθνικά κοινοβούλια δεν μπορούν να παίξουν σωστά το ρόλο τους, αλλά συγκεκριμένες προτάσεις όμως τι θα πρέπει να κάνουμε για να υπάρξει κοινοβουλευτικός δημοκρατικός έλεγχος. Δεν βρήκα πολλά στη μελέτη σας γι' αυτό. Έχετε τίποτα άλλο μπορείτε να μας πείτε. Τέταρτον, που δεν έχει να κάνει απευθείας με τη μελέτη σας, αλλά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο γενικότερα. Εμείς, οι ευρωβουλευτές, λάβαμε μια ανοιχτή επιστολή από το δίκτυο κατά του εμπορίου όπλων και λέγεται ότι οι εμπειρογνώμονες ε, που θα είναι στην Ηθική Επιτροπή, στην Επιτροπή Διοντολογίας για την, ε, τις πωλήσει Ευρωπαϊκού Αμυντικού Εξοπλισμού, δεν είναι γνωστό ποιοι θα είναι. Μήπω θα έπρεπε να εκφράσουμε γνώμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει γνώμη για το ποιοι θα πρέπει να είναι σε αυτήν την Επιτροπή. Και μήπω θα έπρεπε ακριβώ στον καθορισμό αυτών των εμπειρογνωμόνων να έχει λόγο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Πολύ διορατική. Βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει αυτή η διακυβερνητική διάσταση, γιατί η άμυνα είναι μία από τις κύριες ε, αρμοδιότητες των κρατών μελών, ακόμη και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Όταν ε, ομόφωνα αποφασίζεται να ξεκινήσει μια επιχείρηση, αυτό εξαρτάται μετά από εθνικές πολιτικές αποφάσεις να δοθούν συγκεκριμένες δυνατότητες για την ε, υλοποίηση αυτής της αποστολής. Αυτό ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα η διαδικασία στα εθνικά κοινοβούλια για τον έλεγχο, όπως λέει και η μελέτη, είναι πολύ διαφορετικές. Στη χώρα μου, την Εστονία, Έχουμε την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία ασχολείται με την έγκριση των ε, εντολών των Υπουργών για τις συναντήσεις ε, του Συμβουλίου των Υπουργών. Και μετά ο έλεγχος είναι εάν ε, ακολούθησε την εντολή, συμμορφώθηκε με αυτή την εντολή η κυβέρνηση. Δεν, ελέγχει λοιπόν κανείς εάν υπήρξε κατόπιν εφαρμογή των αποφάσεων. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Προπολογισμών, η Επιτροπή για την Εθνική Άμυνα, όταν εξετάζουν τις αμυντικές δαπάνες της χώρας μου, ε, εξετάζουν τα μακροχρόνια σχέδια, το ρόλο μας στο ΝΑΤΟ και στα πλαίσια των στόχων της Ένωσης για την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Οπότε αναφέρατε κάποιους στόχους για να γίνεται ο έλεγχος σε βράχη και πρόθεσμο επίπεδο. Εάν αυξάνεται, για παράδειγμα, η ανταγωνιστικότητα της ε, ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Μα είναι διάμεση στόχη αυτή, γιατί αν έχουμε πιο ανταγωνιστική αμυντική βιομηχανία, θα συμβάλλουμε περισσότερο στις εθνικές δυνατότητες των κρατών μελών. Πολύ λίγα προγράμματα είναι πραγματικά προγράμματα που ευνοούν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, για παράδειγμα οι δορυφόροι. Πολύ λίγα άλλα. Και δεν ξέρω αν συμβάλλουν στις εθνικές δυνατότητες ή αν αντιμετωπίζουν τα κενά, τις ανεπάρκειες των συλλογικών δυνατοτήτων. Όλα αυτά κυρίως εξαρτώνται από εθνικές αποφάσεις. Αν δηλαδή δώσουν πρόσβαση στις εθνικές τους δυνατότητες στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έπρεπε να έχουμε κάπω ευρύτερου στόχου για μια ένωση που να έχει περισσότερε στρατιωτικέ δυνατότητε. Όχι να μιλάμε μόνο για ανταγωνιστικότητα της ε, αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο με την στενότερη έννοια. Ο λόγος στον κύριο να μας απαντήσει στα ερωτήματά μας. Thank uh, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα σημεία και να επιχειρήσω κάπως να γκρουπάρω τις απαντήσεις μου. Συγγνώμη αν θα απαντήσω με τη σειρά που υποβλήθηκαν οι ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να τις ε, συνοψίσω λοιπόν. Λοιπόν, ε, πώς μπλέκονται τα εθνικά κοινοβούλια. Βεβαίως, πρέπει να τονίσω ότι είναι σημαντικό και το θέμα της κυριαρχίας και ο ρόλος των κυβερνήσεων. Και η ΠΕΣΚΟ, η μόνιμη Διατρομένη συνεργασία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας δεν αφαιρούν ε, κυριαρχία από τα κράτη-μέλη. Αυτό που κάνουν είναι δίνουν μια νέα δυνατότητα συνεργασίας για να αναπτυχθούν δυνατότητες, για να υπάρξουν προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία θα αυξήσουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, και θα αυτό αυτό που είπατε, αλλά και τη δυνατότητα και τη Ένωση συνολικά. Βεβαίως, τι δυνατότητε, θα τις κατέχουν πάντα τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν πότε θα ξεκινήσουν αποστολές, επιχειρήσεις. Αλλά θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτές τι δυνατότητε στο μέλλον. Φυσικά, τονίζουμε ότι όλα αυτά έχουν και εθνική διάσταση. Τώρα για το ρόλο της Επιτροπής και άλλων θεσμών, όπως ο Οργανισμός Άμυνας, δεν βλέπω αντιφάσεις εδώ. Ενισχύουμε τις δυνατότητες της Ένωσης συνολικά, μειώνουμε την σημασία ενός ε, παλιού προγράμματος, επικάλυψη, διπλό κόστος, το οποίο έχει επιπτώσει και στη βιομηχανία, αλλά έχει επιπτώσει και για τις δυνατότητές μας. Σωστό λοιπόν είναι το Ταμείο να προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Εγώ δεν βλέπω αντιφάσεις εδώ. Αξιοσημείωτες. Τώρα, τι θα πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο για να αυξήσει τη δυνατότητά του να παίξει ρόλο, δηλαδή να αποκτήσει περισσότερη εμπειρογνωμοσύνη. Υπάρχει ένα ευρύτερο πολιτικό θέμα, θα έλεγα, από πλευρά ελέγχου και επίβλεψη. Τι θέλει η Ένωση, που θέλει να πάει ω ομάδα κρατών μελών και θεσμών στο μέλλον. Αυτό είναι σαφές. Λέμε ότι πρέπει να παίζει ρόλο η Ένωση, αλλά παρόλα αυτά ίσω να μην είναι και τόσο σαφές. Δεν ξέρουμε τι ρόλο από στρατιωτική και διπλωματική άποψη θέλουμε να έχει η Ένωση στον κόσμο. Είναι μια πολύ σκόπιμη συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Άμυνα, τι θέλουμε να γίνει και πόσα θα επενδύσουμε. Το δεύτερο πολύ πιο τεχνικό θέμα, σε άλλο επίπεδο, είναι ε, ο έλεγχος και επίβλεψη συγκεκριμένων προγραμμάτων. Βεβαίως. Εδώ θα μας βοηθήσει και πώς γίνεται ο έλεγχος των εθνικών προγραμμάτων. Πώς παρεμβαίνουν τα κοινοβούλια όταν αναπτύσσουν δυνατότητες στα κράτη-μέλη. Σε ποια φάση. Συνεχώς, στο τέλος, στην αρχή, όπως φαίνεται ότι γίνεται σε κάποια κράτη-μέλη. Εγώ δεν έχω απάντηση για το πώς θα πρέπει να κάνετε σε αυτόν τον έλεγχο. Αυτό που λέω είναι ότι ξεκινάμε από ένα πιο θεμελιώδες θέμα. Υπάρχει θέμα έλλειψης τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης. Στο σώμα σας αλλά και γενικότερα στους θεσμούς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Πώς θα το αντιμετωπίσετε. Στη μελέτη μου προτείνω κάποια θέματα για την Κόζακ και την διακοινωνιστική διάσκεψη δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Πρέπει να είναι πολύ πιο εξειδικευμένε οι συζητήσει του για τα θέματα αυτά στα εθνικά κοινοβούλια. Ανάλογα με το ποια επιτροπή είναι αρμόδια, γιατί ανά χώρα είναι διαφορετικές αυτές οι επιτροπές, όχι πάντα οι ίδιες, από χώρα σε χώρα, ακόμη και σε αυτές τι συζητήσει. Τι γίνεται, ενημερώνονται από το Υπουργείο Άμυνας και μετά περνάνε σε άλλα θέματα δεν είναι μια στρατηγική συζήτηση για το ποιο είναι το κόστος κτλ. Είναι απλώς μια ενημέρωση. Και ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Οι εθνικές κυβερνήσεις πραγματικά έχουν κάθε συμφέρον. Λέμε ότι γίνεται για να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα. Αλλά θέλουμε ακριβώς να ευνοήσουμε και τις μικρομεσαίες και τις εταιρείε μεσαίας κεφαλαιοποίησης. εθνικά κοινοβούλια σε πολλά κράτη-μέλη ενδιαφέρονται πραγματικά το Ταμείο να επιτυγχάνει τους στόχους του. Δεν έχω, δεν έχω φόρμουλες, δεν έχω ολοκληρωμένες λύσεις. Εγώ απλώς επισημαίνω τα προβλήματα. Και προβλήματα είναι ποια δυνατότητα έχετε. Πέρα από μια γενική συζήτηση, πραγματικά να επιβλέψετε, να ελέγξετε τη λειτουργία του Ταμείου. το γεγονό ότι είναι περιορισμένη πόροι του τώρα, του ταμείου αυτού. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τις, ε, από τις ε, εταιρείε μελετών, από τις, ε, τους ομίλους μελετών. Πολλοί λένε, χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα, λένε, αλλά κοιτάξτε, το, το θέμα δεν είναι μόνο η πόρη. το θέμα είναι και η διαδικασία. Το Ταμείο Άμυνας είναι ένα νέος τρόπος συνεργασίας. Να τονιστεί αυτό. Σημαντική η πρικοδότησή του, αλλά πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία και ίσως να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αλλάξουν νοοτροπία. Τα κράτη-μέλη έχουν κάθε συμφέρον φυσικά να διασφαλίσουν ότι θα λειτουργήσει το Ταμείο. Θα πάει καλά. Και το τονίζω. Να μην ξεχνάμε ότι αναφέρονται 13 δις βεβαίως, αλλά κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον είναι οι δυνατότητες μόχλευσης για να βοηθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Να μην το ξεχνάμε. Πολιτική πορεία τη Ένωση στον τομέα τη άμυνα. Τώρα. Έγιναν και κάποιε άλλες ερωτήσει, δεν ξέρω αν έχω απαντήσει. Σωστό, ισχύει ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ρόλο κλειδί να παίξουν. Βεβαίω. Να μην ξεχνάμε ότι τα διάφορα εθνικά κοινοβούλια αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο το θέμα και της Ευρωπαϊκής Άμυνας και της Άμυνας γενικότερα. Δεν έχω συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς πρέπει να οργανώσετε εσείς αυτό τον έλεγχο. Τι άλλο. Α, ναι. υπόθηκε το σχόλιο για το ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι φορεί ε, ποιε επιχειρήσει τα κράτη-μέλη, αλλά και για τον κλάδο. Είναι ενδιαφέρον. Ποτέ δεν χρειάστηκε να συνεργαστούν με αυτόν τον τρόπο στο παρελθόν. Άρα έχουν και αυτές πολλά να μάθουν. Να σταματήσω εδώ. Μα πάρα πολύ. Μία ακόμα Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μία διευκρίνηση ήθελα να ζητήσω. Στη συζήτηση που είχαμε, όταν εγώ μίλησα για το περιορισμένο ποσό που διατίθεται μέσω του Ταμείου, είναι σημαντικές διαδικασίες, αλλά αυτό που λέτε με καλύπτει, συμφωνεί με αυτό που είπα. Δηλαδή, το Ταμείο Αμήνης δεν θα χρηματοδοτήσει από μόνο του κανένα άργο έργο αμυντικών εξοπλισμών. Εξ ολοκλήρου. Το Ταμείο θα συνεισφέρει, θα υποστηρίξει διάφορα έργα, αλλά θα συνεισφέρει σε ένα μικρό μέρος και σε έργα που θα είναι συνεργασίες μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να μοχλεύσει, ώστε να βοηθήσει. Και εκεί θα πρέπει να ε, ασκήσουμε και τον κοινωνικό μας ε, έλεγχο, αλλά ε, λυπάμαι, αλλά αυτό σημαίνει ότι και ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το EDF ε, θα ελέγξει το 25% μια συνεισφορά σε ένα ευρύτερο έργο. Και εκεί για τα υπόλοιπα θα μιλούμε για εθνικά κονδύλια. Συνεργασίες δηλαδή διακρατικής μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποια είναι και τα μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας για να ασκήσουμε ποιον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δηλαδή είναι ακόμα πιο σχετική η σημασία του ελέγχου που θα ασκήσουμε σε σχέση μάλιστα με αυτή που καλούνται να ασκήσουν τα εθνικά κοινοβούλια. No, I don't dissent. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συμμετοχή σας. Έληξε συνεδρίαση μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς ε, να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος ε, ανέλαβε τα ενία της Προεδρίας ε, την πρώτη ώρα της συνεδρίασης, να καλωσορίσω εξ ονόματος όλων την Ελισαμπέτα Μπιενκόφσκα, Επίτροπο Αρμόδια Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μια Επίτροπο η οποία ε, συνέβαλε για να αλλάξει ο τρόπος ε, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με τα θέματα της ε, άμυνας. Μπορούμε να το πούμε εδώ στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ. Όταν αναλάβατε τη θητεία σας το 2014, λάβατε μια επιστολή για την αποστολή σας από τον πρόεδρο Γιούνκερ, στην οποία υπήρχε η παράγραφος, στην οποία θα διαβάσω τα αγγλικά, ενθαρρύνοντας τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν περισσότερες συνέργειες και μεγαλύτερη συνεργασία στις ο διαγωνισμός της άμυνας στι αμυντικέ ε, προμήθειε, ε, προκειμένου να αποφύγουμε επανάληψη των εθνικών προγραμμάτων και να έχουμε πόρου αντίστοιχου με του ε, στόχου εξωτερική μα πολιτική. Νομίζω ότι σα έδωσε τη μέγιστη δυνατή εντολή και φυσικά τα θέματα της άμενας πλουτίστηκαν πάρα πολύ, κυρίως μετά το 2016 και ξεκίνησε η συνολική στρατηγική προβλέπεται η σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την άμυνα μεταξύ των σχεδίων της άμυνας και ο στόχος είναι να υπάρχει πιο αποτελεσματική ε, χρήση των κονδυλίων, στις δυνατότητες άμυνας ε, που προσπαθούμε να στήσουμε σε κοινό επίπεδο, να ενισχύσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και να έχουμε και ε, ανταγωνιστική και καινοτόμο βιομηχανία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει λοιπόν και ένα δημοσιονομικό εργαλείο προκειμένου να διαμορφώσει την βιομηχανία της άμυνας των κρατών μελών της. Το 2017 είχε πολύ σημαντικές προόδους για τα θέματα της καινοτομίας και της στήριξη τη ανταγωνιστικότητας τη βιομηχανία βιομηχανίας της άμυνας ε, με την ε, ε, διαρθρωμένη δομή συνεργασίας και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το EDIDP. Ε, βέβαια, ακόμα πρέπει να οριστικοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Οι νομοθέτες ε, κατέληξαν σε μια μερική συμφωνία για την πρόταση κανονισμού του Ταμείου στις 19 Φεβρουαρίου, που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 17 Απριλίου του 2019, αλλά υπάρχουν ακόμα δύο σημεία στα οποία δεν έχουν ε, ε, διευκρινιστεί. Το ποσό του Ταμείου και τη συμμετοχή των τρίτων χωρών. Ε, ξέρουμε ότι το τελευταίο αφορά περιορισμένο άνοιγμα του Ταμείου σε επιχειρήσεις των συνδεδεμένων χωρών, κυρίως ε, το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Και τα μέλη της Επιτροπής μας ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη δική σας ανάλυση για αυτές τις προκλήσεις και για τον απολογισμό που θα μας κάνετε για τις ε, προόδους που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Έχετε το λόγο κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εδώ μαζί σας για τη συμβολή και το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποχωρεί όσον αφορά την συνεργασία σε θέματα άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι υπερβήκαμε αυτά τα οποία περιλάμβανε η επιστολή του Πρόεδρου Γιούνκερ. Ε, πλέον δεν αφορά μόνο τις δημόσιες προμήθειες το θέμα αυτό. Έχουμε κάνει ένα άλμα ε, και ε, προωθούμε την συνεργασία για την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νέο επίπεδο. Να σας υπενθυμίσω ότι ξεκίνησε το 2014, ακόμα και από πριν δηλαδή αναλάβει καθήκοντα η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη στις προσπάθειες μετά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της υποεπιτροπής σας, για πρώτη φορά έχουμε στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό κονδύλια ειδικά για την έρευνα ε, στον τομέα της άμυνας. Αυτή ήταν η αρχή. Ε, ήταν μια πιλωτική δράση για την έρευνα και την άμυνα. Έκτοτε έχουν συμβεί πάρα πολλά. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κράτος μέλος ε, το οποίο ε, μπορεί να αντιμετωπίσει τεράστιες ε, σύνθετες ε, προκλήσεις από μόνο του. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη η οποία θα παρέχει ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα σταδιακά θα εξασφαλίζει και τη δική της την προστασία το να δημιουργήσουμε μία αξιόπιστη ε, ένωση άμυνας ε, δεν είναι κάτι το οποίο αντιβαίνει στα όσα κάνει το ΝΑΤΟ. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα σχεδιάσουμε τα προγράμματα και αν οργανωθούμε σε θέματα άμυνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να γίνει πιο αξιόπιστος εταίρος για ε, κάθε, μία, κάθε έναν από τους συμμάχους μας. προχωρούμε με τα θέματα της άμυνας, ξεκινήσαμε με την έρευνα, και τις προπαρασκευαστικές δράσεις για την έρευνα, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια ε, στην άμυνα επιτύχαμε πολύ περισσότερα από ότι τα τελευταία 60 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έναρξη του ΠΕΣΚΟ, της ε, διαρθρωμένης συνεργασίας ε, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Θα επανέλθω εντός ολίγου από αυτού. Να σας υπενθυμίσω ότι σε κάθε στάδιο των εργασιών μας προσέξαμε πάρα πολύ ώστε να ενισχύσουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ. Αυτός ε, ήταν ε, ο βασικός μας στόχος. Μετά από δύο κοινέ ε, δηλώσεις, η σχέση πλέον είναι επιχειρησιακή σε αρκετές διαστάσεις. Στρατιωτική κινητικότητα, υβριδικά ζητήματα, ασφάλεια. και φυσικά εμείς θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το ρόλο μας ως πάροχος ασφάλειας αν εντατικοποιήσουμε και ενισχύσουμε ανταγωνιστικές και καινοτόμες ε, επιχειρήσεις ε, στον τομέα της άμυνας. Γι' αυτό έρχομαι και εγώ εδώ με το δικό μου το χαρτοφυλάκιο. Ξεκινάμε λοιπόν με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητές μας ε, και της βάσης μας σε καινοτομία στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Αυτό που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε ακόμα είναι ότι έχουμε ένα κατακαιρματισμένο πεδίο στην άμυνα με χαμηλές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Το Δεκέμβριο του 2016 ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, ανακοίνωσε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για να ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη σε θέματα άμυνας και έκτοτε χάρη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη στήριξή του ξεκίνησαν δύο προγράμματα μικρής κλίμακας, ε, τα οποία είναι ήδη ε, σε εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν την ε, έρευνα για το Κοινοβούλιο έχουμε 90 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν ε, από τις τελευταίες ε, διαδικασίες διαγωνισμών. Έχουμε ακόμα 7 προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και ελπίζουμε ακόμα σε, να έχουμε 18 ερευνητικά προγράμματα στα μέσα του επόμενου έτους. Και επίσης υπάρχει και το Ocean 2020, πάντα το αναφέρω αυτό το πρόγραμμα, διότι έρχεται να συγχωνεύσει όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε. Σε αυτό το ε, σχέδιο έχουμε 42 οντότητες από όλη την Ευρώπη και αποτελεί παράδειγμα πραγματική ευρωπαϊκής συνεργασίας. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο μικρότερο πρόγραμμα, ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι υποδοκιμή, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης για την Άνουνα. Έχουμε 500 εκατομμύρια ευρώ εδώ, το οποίο ε, έχει ξεκινήσει την υλοποίησή του και εδώ έχουμε το πρώτο ε, πρόγραμμα άμυνας που ενέκριναν οι συνομοθέτες σε ένα χρόνο ε, και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό ότι έγινε τόσο γρήγορα η έγκριση και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει με ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και μέσω του μοντέλου συγχρηματοδότησης ένα ε, κοινό βιομηχανικό πρόγραμμα για την άμυνα. Έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο πιλωτικά προγράμματα όπως τα αποκαλούμε. Μέσω αυτού του προγράμματος, το πρόγραμμα της βιομηχανικής ανάπτυξης, ο κλάδος μπόρεσε να υποβάλει προτάσεις η προθεσμία έληξε την ε, προηγούμενη Παρασκευή, 20 ε, Σεπτεμβρίου και του χρόνου θα έχουμε έναν επόμενο γύρο. Και εδώ έχουμε τις εξής προτεραιότητες. 80 εκατομμύρια ευρώ για να υπάρχει επιχειρησιακή προστασία και κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων, 180 εκατομμύρια για πληροφορίες, ε, συντορισμό ασφάλειας και κυβερνοασφάλεια, 400 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια, συγγνώμη, για να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και 27 εκατομμύρια για προγράμματα που καλύπτουν καινοτόμε ε, τεχνολογίες και εδώ περιλαμβάνουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί κάθε στάδιο των προγραμμάτων ε, επισημαίνει και την παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης ε, συγχρηματοδοτούνται και δύο σημαντικά προγράμματα PESCO. Θα τα αναφέρω αλλά θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνοχή στη διάφορα παρακλάδια της εργασίας μας ε, και αυτά τα οποία προτείνει η Πατή Εκπρόσωπος, αλλά και το βιομηχανικό σκέλος το οποίο μας απασχολεί. Αυτά τα δύο προγράμματα ΠΕΣΚΟ λοιπόν είναι η ανάπτυξη των Eurodrones 100 ε, εκατομμύρια ευρώ και το πρόγραμμα ESOR 37 εκατομμύρια για τη διαλειτουργική και ασφαλή συστήματα άμυνας και συνεργασίας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πολύ σημαντικό σκέλος του προπολογισμού θα ε, αφορά διασυνοριακή συνεργασία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό είναι να ανοίξουμε και την αλυσίδα αξία του κλάδου και ε, σε νέους συμμετέχοντες. Όπως σας είπα όμως αυτά είναι μόνο πιλωτικά προγράμματα. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο έχει προτείνει 13 δις ευρώ τα οποία θα είναι για το πλήρες Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας συν 65 ε, δισεκατομμύρια για να υποστηρίξουμε τη στρατιωτική κινητικότητα. Χάρη στην πολιτική βούληση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μπορέσαμε λοιπόν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο Καταλήξαμε σε συμφωνία για τα βασικά στοιχεία του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα. Εγώ συμμετείχα προσωπικά και διεξήγαγα τι διαπραγματεύσει και μπορώ να σα επιβεβαιώσω ότι υπήρχαν πολλά εξαιρετικά σημαντικά σημεία ε, τα οποία επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελήφθησαν υπόψη. Να αναφέρω εδώ ε, τέσσερα πολύ σημαντικά στοιχεία. Καταρχάς, εξασφαλίσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ε, έχει συνοχή με πρωτοβουλίες άμυνας ε, υπό την πολιτική εκκλησία της υπάτηση εκπροσώπου. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, γνωρίζουμε και τα ειδοντολογικά ζητήματα. Έγινε πολύ μακρά συζήτηση στον τριμερή διάλογο επ' αυτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να ε, δημοσιεύσει δεοντολογικό ε, οδηγό, αν θέλετε. Επίσης, έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα το γεγονός ότι οι δράσεις που αφορούν ε, συστήματα αυτόνομων όπλων δεν θα χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Δεν υπάρχει δηλαδή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για αυτά. Και ένα τέταρτο, ο κανονισμός ε, επικεντρώνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε τεχνολογίες εχμής. Το 80% του προπολογισμού αφορά αυτά τα θέματα. Υπάρχουν ακόμα δύο εκκρεμότητες. Το πρώτο είναι πρωτίστως ο προπολογισμό, που είναι τμήμα των συνολικών διαπραγματεύσεων για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και εδώ πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω τη μόνιμη και συνεχή υποστήριξή σας γιατί τη χρειαζόμαστε. Χάρη στα κίνητρα που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον προπολογισμό, τα οποία είναι ελάχιστα σε σχέση με την κλίμακα και τον όγκο του κλάδου, μπορέσαμε να σχεδιάσουμε την αρχή της ε, πολιτικής άμυνας ε, της Ευρώπης δεν είναι μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί μία ή δύο χώρε, αλλά είναι μια πολιτική η οποία υποστηρίζεται από όλα τα κράτη-μέλη και έχουμε και το άκουσα ε, και από όλου ε, τεράστια υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαφορετική προσέγγιση που υπάρχει από κάθε χώρα στην άμυνα. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό. Αυτό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα θέματα που αποσχολούσαν το χαρτοφυλάκιό μου είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει υποστήριξη των 28 κρατών μελών. Θα ήθελα εδώ να είμαι σαφής, γιατί αυτά τα θέματα πάντα ε, ανακύπτουν και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνάς δεν είναι ε, εργαλείο προστατευτικότητας. Κάποιοι προσπαθούν να τα παρουσιάσουν ω τέτοιο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχαμε αυτή την πρόθεση, δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας και ευθύ εξ αρχή ε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με όλους μας τους εταίρους ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπα και στην αρχή, οργανώνει ακριβώς το νομικό πλαίσιο για τη συμμετοχή τρίτων χωρών επιχειρήσεων από τρίτες χώρες, ε, όλες επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μπορεί να μην είναι υπό τον άμεσο ευρωπαϊκό έλεγχο. Δεν απορρίπτεται δηλαδή κανένας, ε, αντιθέτως, το Ταμείο δεν ε, παρακολεί τη συνεργασία με τους εταίρους μας, ούτε ε, αντιβαίνει στους ε, κανόνες περί μειοδοτικών διαγωνισμών της Ευρώπης, ίσα ίσα Επιμένω αυτό, είναι πολύ πιο ανοιχτό στις αγορές. Οι ευρωπαϊκές αγορές είναι πιο ανοιχτές σε σχέση με τις αγορές ε, κάποιων από τους στενότερους συμμάχους μας. Δεν θα αντικαταστήσουμε Κανέναν ούτε θα εμποδίσουμε τέτοια προγράμματα στο μέλλον. Δεν πρόκειται να επηρεάσει τα δικαιώματα εξαγωγών των κρατών μελών. Αυτά είναι δικαιώματα των κρατών μελών. Και τι προσθέτει αυτό το ταμείο. Είναι η συνεργασία. Αυτή είναι η προστεθέμενη αξία. Δεν εμποδίζει τίποτα, δεν αντικαθιστά τίποτα, απλώς διευκολύνει την ευρωπαϊκή συνεργασία. Και δεν θα οδηγήσει σε λιγότερη διαλειτουργικότητα. Ο στόχος μας από την αρχή ήταν να μειωθούν οι επικαλύψεις, να αυξηθεί η διαλειτουργικότητα και με τον ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η συμμετοχή υπάρχει η επιλεξιμότητα για τους ε, πόρους του προϋποθέτουν την τήρηση κάποιων κριτηρίων που είναι ο στόχος μας. Πρώτα απ' όλα να διατηρούνται τα συμφέροντα ασφαλείας της ε, Ένωσης, οποιαδήποτε εταιρεία, οποιαδήποτε επιχείρηση, φορέας που θέλει να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο, πρέπει να σέβεται αυτά τα κριτήρια, τα οποία είναι παρόμοια σε αυτά, προς αυτά που πρέπει να τηρούν οι δικές μας επιχειρήσεις όταν πρέπει να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς σε άλλες χώρες. Φυσικά σε στενή συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Άρα περισσότερη συνεργασία στην Ευρώπη και αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων. Αυτός είναι ο γενικός μας στόχος. Έτσι θα μπορέσουμε να παίξουμε ένα ισχυρότερο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή και να αναλάβουμε το τμήμα της ευθύνης και του βάρους των αμυντικών προσπαθειών που μας αναλογεί όπως μας καλούνε κάποιοι εταίροι μας. Θα μας επιτρέπει να συμβάλλουμε καλύτερα στον ΝΑΤΟ, περισσότερη διαλειτουργικότητα και τελευταίας γενιάς εξοπλισμούς. Θέλουμε να μπορέσουμε να αλλάξουμε εκ την κατάσταση. Έχουμε ένα μοντέλο συγχρηματοδότησης μέσω του οποίου μαζί και με κάποια μπόνους που μπορεί να λάβει κανείς θέλουμε να ευνοήσουμε, να προωθήσουμε τη συνεργασία των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να προωθήσουμε και τις αλυσίδες αξίας. Και θέλουμε να αυξήσουμε και τις δυνατότητες άμυνας μέσω διαστήματος. Ξέρω ότι θα τα συζητήσετε και αύριο. Υπάρχει σαφή σύνδεση της χρήσης του διαστήματος και της ε, άμυνας. Θέλουμε ε, επικερδείς συνεργασίες μέσω της ΠΕΣΚΟ και του Ταμείου Άμυνας. Τα προγράμματα ΠΕΣΚΟ θα έχουν υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Κοιτάξτε, είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά, το τονίζω. Πραγματικά δημιουργούμε καλές προϋποθέσεις για την επόμενη Επιτροπή. Έχουμε δύο πιλωτικά προγράμματα που είναι δοκιμές ας πούμε για την πλήρη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου και θεωρώ ότι οι στόχοι μας είναι όντως ρεαλιστική. Χρειάζεται βούληση, αποφασιστικότητα και ε, σωστή τήρηση των διαδικασιών. Για υποβολή αιτήσεων, για παράδειγμα. Πιστεύω ότι η Επιτροπή σα για άλλη μια φορά θα μα στηρίξει, γιατί χρειάζεται μια λίγο καλύτερα, περισσότερη προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για κάποιε διατάξει που εκκρεμούν του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνα. Άρα βασίζομαι σε εσά, είναι κάτι που είναι σημαντικό για την αμυντική μα βιομηχανία, που δημιουργεί και πολλέ θέσει εργασία και σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω πρώτα το λόγο στους ε, συντονιστές που ζήτησαν το λόγο. Πρώτος ο Αγνόντα Οζόν για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Είναι μάλλον η τελευταία φορά που είστε στην ε, υποεπιτροπή μας από πλευρά της πολιτικής ομάδας. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την εργασία που επιτελέσατε, η οποία είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Το είπατε κι εσείς βέβαια. Το είπε και η Πρόεδρος. Πολλά ακόμη πρέπει να ρυθμιστούν για αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που είναι φιλόδοξο και καλοδεχούμενο. Εντάξει, δεν θα το χαρακτήριζα και εκβάθρον ανατροπή της κατάστασης. Ε, καταλαβαίνω ότι πρέπει να τα πείτε αυτά. Υπάρχουν ε, κάποιες αδυναμίες ακόμη, ατέλειες του όλου εγχειρήματο. Πρέπει να προσέξουμε για να μην ξεφύγουμε. Υπάρχουν ε, πολύ σοβαρά θέματα. Το θέμα των τρίτων χωρών είναι πολύ περίπλοκο. Καλά κάνατε που υπενθυμίσατε ότι οι τάσεις προστατευτισμού είναι ιδιαίτερα άδικες. Μάλλον οι επιθέσεις που μας κάνουν ότι, ασκούμε προστατευτισμό είναι άδικες. Και κάτι άλλο που μπορούμε να τονίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά είναι ότι κάποιοι σύμμαχοί μας είναι πολύ πιο προστατευτική από εμά. Εγώ νομίζω ότι είμαστε εμεί υπερβολικά ανοιχτοί. Ελπίζω στην επόμενη θητεία να μπορέσουμε να συζητήσουμε και για κάποια θέματα που τα αποφεύγουμε όπω ο διάλογο στο Λιβάνι. Δηλαδή, αν εφαρμόζουμε ή όχι την κοινωνική προτίμηση. Ενώ μα επιτίθεται. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την εργασία που επιτελέσατε, αλλά τώρα που ξεκινάει η νέα επιτροπή, όπω είπα και στην προηγούμενη συζήτηση, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και εδώ ακριβώς είναι αυτό το οποίο επιτύχατε σημαντικό. Καταφέρατε αυτό το πρόγραμμα να προχωρήσει με πολύ περισσότερη πρωτοτυπία από ό,τι συνήθως περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ ευελιξία, πολύ ταπεινοφροσύνη. Και παρόλα αυτά καταφέρατε με πολύ ευέλικτο τρόπο, με τρόπο που αντιδρά στα γεγονότα, να καταφέρετε να συγκεντρώσετε γύρω από το τραπέζι και να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη και οι επιχειρήσεις. Και αυτή η αλχημία με την οποία προωθείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι καταπληκτική. Εάν υπάρξουν παραφωνίες μεταξύ των κύριων συμμετεχόντων υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Εάν οι επιχειρήσεις ή τα κράτη-μέλη θεωρήσουν ότι η βαριά γραφειοκρατία της Κομισιόν, με που το λέω έτσι, θα έχει το πάνω χέρι, τότε μπορεί να έχουμε απώλειες. Ελπίζω λοιπόν οι διάδοχοί σας να έχουν την ίδια προσέγγιση. Η αμυντική βιομηχανία δεν είναι μόνο βιομηχανία. Η αμυντική βιομηχανία έχει να κάνει με θέματα κυριαρχίας, ε, λειτουργικά, επιχειρησιακά, εμπορικά είναι πραγματικά ένας ιδιαίτερος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας. Όταν βλέπω λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί μια, ε, θα δημιουργηθεί μια πολύ συνήθις δομή μέσω μιας Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία αυτής της μηχανίας, θεωρώ ότι αυτή η εξομάλυση του τρόπου λειτουργίας μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων άμυνας τα καταφέρατε, ελπίζω και οι διάδοχοί σας να το επιτύχουν. Ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι οι εντυπώσεις σας, ποιες συμβουλές θα είχατε να δώσετε σε αυτούς που θα, θα σας διαδεχτούν. Άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για όσα κάνατε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και εγώ είχα την αίσθηση αυτή και κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει καλύτερα από μένα πόσο <laughs> η υπερβολική γραφειοκρατική δομή γεννάει τέρατα, για να το πω έτσι. Ε, εμείς τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε προετοιμαστεί για την διάκριση αυτής της αρμοδιότητας της συγκεκριμένης. Ε, για μένα ήταν σαφές εδώ και μήνες ότι τόσο σημαντικά τμήματα του χαρτοφυλακίου όσο το διάστημα και η άμυνα και που αυξάνονται και μεγεθύνονται συνέχεια παρότι δεν είναι τεράστια κονδύλια σε σχέση με τον κλάδο αλλά είχαμε ξεκινήσει από το μηδέν από την άλλη. Ε, ελπίζω λοιπόν και πιστεύω ότι μέσω αυτής της φάσης δοκιμών των πιλωτικών που κάναμε καθότι ήμουν σε πολύ στενή επαφή και το έλεγα ανοιχτά. Με τα κρατημέλη, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, καθότι δεν είχαμε και ακόμα δεν έχουμε επαρκή εμπειρογνωμοσύνη εντό Κομισιόν, η νέα γαμαδέλτα θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να αντλήσει κι άλλη εμπειρογνωμοσύνη από τα κρατη Και σε διάφορες περιπτώσεις είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους υποβάλλοντες ε, για τα έργα, οι οποίοι είχαν διάφορες, διάφορα ενδιαφέροντα και διάφορες ερωτήσεις. Αλλά η πρώτη απάντηση ήταν τα ενωσιακά κονδύλια έχουν δυσκολίες. Πάντα. Δυστυχώς. Είναι πόροι, χρήματα που δίδονται. Και επομένως ε, πρέπει να έχουν κάποιες εγγύησεις. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι η όλη διαδικασία ε, πρέπει να είναι και τελείως εχθρική προς ε, τους ενδιαφερομένους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η φάση δοκιμών και ερευνητικά και επί του δυναμικού προσφέρει στην Γενική Διεύθυνση, στις υπηρεσίες ε, και στην μελλοντική σύνδεση, στην επερχόμενη σύνδεση κομισιών, την απαραίτητη γνώση, εμπειρία να μην μας ξεπερνάει αυτό το γραφειοκρατικό οικοδόμημα. Χρειάζονται κίνητρα. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να το οικοδομήσουμε ως μέσο που θα απευθύνεται προς τις επιχειρήσεις και θα είναι φιλικό προς αυτές. Η ίδια η διεύθυνση θα αναπτυχθεί, το ξαναλέω. Και θα έχουμε και άλλους ανθρώπους και άλλους συνεργάτες. Ο κύριος Ριβιέχ, ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αναφερθήκατε σε απαραίτητες συνεργασίες πρέπει να έχουμε με τη βιομηχανία και βεβαίως στο αμυντικό πεδίο είναι απολύτω απαραίτητο. Αλλά εδώ είναι που θα διαφωνούσα ελαφρώς με τη δική σας ανάλυση εσείς εξηγήσετε με μεγάλη διαφάνεια την φιλοσοφία, την πολιτική που ε, κινούσε τις προσπάθειές σας ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πλέον παίκτη στο επίπεδο των αμυντικών εξοπλισμών και υπέρ της κυριαρχίας και των κρατών μελών. Ακολουθώντας λοιπόν μία οδό η οποία οδηγεί στην συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενεργητική την ενεργό συμμετοχή στα αμυντικά θέματα. Τώρα, για τι συνεργασίε. έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ε, διμερών συνεργασιών αναγκάζοντας να είναι τουλάχιστον τρεις χώρες για παράδειγμα όταν λέμε για ένα έργο για να συνεργαστούν όλα αυτά τα χρήματα οι πόροι οι ερευνητικοί ε, διοχετεύονται σε συνεργασίες που ξαναγκάζουν τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν σε ένα πράγμα το οποίο μπορεί να μην τους ενδιέφερε εάν είχαν την απόλυτη ελευθερία. Επομένως υπάρχει ένας φεντεραλισμό, μια φεντεραλιστική κατεύθυνση σε όλα αυτά, για να το πούμε έτσι. Ε, τώρα, μιλάτε 13 δισεκατομμύρια, ναι, μπορεί να πει κανεί ότι δεν είναι και ένα απίστευτο κονδύλιο, ε, βλέποντας την αγορά και την, των αμυντικών εξοπλισμών, αυτό που εγώ θα έλεγα είναι ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί και να ανακαλύψουμε ότι μπορεί να έχουμε σπατελήσει διάφορους πόρους. Γιατί αυτά τα έργα, τα ερευνητικά, μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένα από τις επιχειρησιακές ανάγκες. Από τα αρχηγεία, τα στρατιωτικά που έχουν ανάγκες συγκεκριμένε αμυντικές. Ίσως είναι αποσυνδεδεμένα κάποια από αυτά τα έργα, λοιπόν, ξαναλέω, από τις επιχειρησιακές ανάγκες των επιτελείων. Πάντως, πράγματι, προχωρήσατε πολύ πέρα από την αρχική εντολή που σας είχε δοθεί, ε, την, ενδεχομένως κάπως στενή. Εγώ σας συγχαίρω ε, και σας ευχαριστώ ε, και θα πρέπει πράγματι να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο στα επόμενα χρόνια με τα θέματα των αμυντικών εξοπλισμών, τα αμυντικά θέματα. Η όπως είπα στην αρχική μου τοποθέτηση, έχουμε την υποστήριξη των 28 κρατών μελών που καθένα από αυτά συνεφώνησε. Ήταν έφορο δηλαδή το πεδίο γιατί όλα τα κράτη-μέλη εξωθούσαν, συνεισέφεραν. Το σημείο κίνησης στο αρχικό βεβαίως ήταν διαφορετικό. Με τι μοιάζει αυτή τη στιγμή ο βιομηχανικός κλάδος. Εμείς έχουμε δεδομένα που μας δείχνουν ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε μέχρι τα και 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως εφόσον έχουμε τέτοιες συνεργασίες. Δεν αποκλείουμε τις διμερείς. Αν κάποιο κράτο μέλο θέλει διμερός να συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο, είναι πολύ ελεύθερο να το κάνει. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να δαπανούμε πιο αποτελεσματικά. Γιατί αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη επενδύουν τους ίδιους πόρους για να αναπτύξουν τα ίδια σχετικά και την ίδια έρευνα. Δηλαδή υπάρχει επικάλυψη. Υπάρχει τεράστιος κατακαιρματισμός, με συγχωρείτε, στην αγορά αυτή τη στιγμή. Είχαμε όμως ενδελεχέστατη ανάλυση της αγοράς με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα και ενδείξεις που μας έδειχναν αυτό το τοπίο. Υπήρχε μια κάποια αντοχή από κάποια κρατημέλη, αλλά από την αρχή μας υποστήριξαν στην προσπάθειά μας αυτή όλα τα κρατημέλη, διότι, ναι, ελάμβαναν πόρους και ξαναλέω, απολύτως δυνατή η διμερή συνεργασία αν θέλετε να ενταχθείτε, να λάβετε πόρους από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, από το EDF και αυτό συνεισφέρει με την εθνική χρηματοδότηση, θα πρέπει να είμαστε σε ένα ευρύτερο πεδίο. Να εχουμε περισσοτερο περισσότερα από δύο κράτη-μέλη, περισσότερες από δύο επιχειρήσεις, να έχουμε και μικρότερες επιχειρήσεις κτλ. Και επαναλαμβάνω διαρκώ. Εάν το ταμείο αυτό έχει μια επιτυχία με 2-3 κράτη-μέλη και 2-3 επιχειρήσεις μόνο, δεν πρόκειται να συνεχίσει επιτυχώς. Θα πρέπει να, να συμμερίζονται τα κράτη-μέλη και οι μικρότερε επιχειρήσεις το αίσθημα ότι είναι επιτυχής η προσπάθεια, ότι είναι αποτελεσματικέ οι επενδύσει οι δαπάνες αυτές σε διάφορα κράτη-μέλη, σε διάφορα επίπεδα και ότι δεν επικαλύπτονται οι προσπάθειες. Δεν δαπανώνται χρήματα για να επιτύχουμε τα ίδια πράγματα σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Ξεκινήσαμε λοιπόν, όπως σας είπα, από μια προοπτική βιομηχανική. Ήταν θέματα με τα οποία είχα ασχοληθεί εγώ, υπό το χαρτοφυλάκιό μου. Και δηλαδή συμπεριλαμβάνοντας την οικονομική διάσταση. Αλλά ιδιαίτερα η ερευνητική διάσταση του προγράμματος πολύ συχνά ε, ε, χειρίζεται τεχνολογίες διτής χρήσεως ή πολλαπλής χρήσεως. Πρόκειται λοιπόν για πρόσφετους πόρους για μια συνεργασία εν ώψη πολύ ευρύτερων γεωπολιτικών στόχων, ναι, αλλά επί τη βάση της οικονομίας, της βιομηχανίας των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ ο κύριος ε, Σούστα. Ευχαριστώ. Ναι, αλλά αυτό με κάνει λίγο διστακτικό. Γιατί ακριβώ ο αμυντικό κλάδο δεν είναι μια συνηθισμένη οικονομική δραστηριότητα. Και μήπω ε, τα κάνουμε τα πράγματα προθύστερα. Αποφασίζουμε ποια οπλικά συστήματα χρειαζόμαστε με βάση μία ανάλυση της πολιτικής ασφάλειας, με βάση μία ανάλυση των απειλών, τι θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο στρατός μας και μετά λέμε τι όπλα χρειαζόμαστε για αυτά. Οπότε δεν είναι δυνατόν δύο, τρία ή πέντε κράτη-μέλη να πούνε θέλουμε αυτά τα οπλικά συστήματα. Και έχουμε κάποιες μικρομεσαίες που λένε ναι, ναι, ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να είναι ουσιώδες κριτήριο αυτό για το τι όπλα θα παραχθούν στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι συνήθις βιομηχανικός κλάδος. Πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Συνήθως δεν λειτουργεί με βάση τους κανόνες της αγοράς. Οι περισσότερες εταιρείες ζουν από τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις. Κανένας δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τις επιδοτήσεις. Αλλά λέμε για λόγους ε, πολιτικής ασφαλείας θέλουμε αυτά τα οπλικά συστήματα. Δεν θα γίνουν όλα αυτά. Και ξέρουμε ότι ναι, μεν θέλουμε περισσότερη συνεργασία, αυτό το χαιρετίζω. Αλλά ακόμη απέχουμε πολύ από μια ενοποιημένη ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτό. Και μετά θέλουμε να ξέρουμε και πώς θα υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Αλλά στα διαφορετικά κράτη-μέλη υπάρχουν πολύ ουσιώδεις διαφορές στον τρόπο άσκησης του δημοκρατικού ελέγχου σε αυτό τον κλάδο. Δεν είναι λοιπόν προθύστερα αυτά που κάνουμε. Πώς θα αποφασίσουμε τι όπλα θα προωθήσουμε και θα επιδοτήσουμε. Ίσως δεν ήμουν σαφής. Γιατί ήταν πολύ τεχνικό, έτσι όπως το παρουσίασα. Στην αρχή έχουμε τις αποφάσεις των κρατών μελών πάντα. Για τις συμπεφωνημένες προτεραιότητες και δυνατότητες. Τα κράτη-μέλη με βάση το CDP, το πρόγραμμα ανάπτυξη δυνατοτήτων και την ΠΕΣΚΟ αποφασίζουν τι προγράμματα, τι δυνατότητες θέλουν. Είναι η δική του απόφαση. Δεν θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιε θα είναι οι προτεραιότητές τους. Οι προτεραιότητε που ανέφερα στα πλαίσια του EDIDP, δηλαδή του προγράμματος ε, ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας, αποφασίζονται από τα κράτη-μέλη. Το πρώτο είναι η επιλογή προγραμμάτων. Και αυτό γίνεται με βάση την υπεράσπιση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Όλα αυτά αποφασίζονται από τα κράτη-μέλη, όχι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο Πέτρας Αουστρεβίχιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω μια άλλη άποψη, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, πολλές τεχνολογίες είναι διπλής χρήσης ε, και αυτό φυσικά μπορεί να οδηγήσει και σε διαφορετικά αποτελέσματα ε, από τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιος θετικός αντίκτυπος ε, στον κλάδο για προγράμματα τα οποία χρηματοδότησε το Ταμείο Άμυνας ε, και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε ποιο βαθμό γίνεται πιο ε, ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία και έχει και καλύτερη θέση ε, μετά από την εμπλοκή και του ε, Ταμείου Άμυνας στο συγκεκριμένο κλάδο. Νομίζω ότι είναι νωρίς να πούμε για τα αποτελέσματα του προγράμματος, διότι μόλις ξεκίνησε ο πρώτος γύρος ε, των ε, προσκλήσεων υποβολής ε, προσφορών για την έρευνα ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και πέρσι ξεκίνησαν τα υπόλοιπα σκέλη για την έρευνα και την ανάπτυξη και τα λοιπά. επομένως είναι τα τελευταία τρία χρόνια των νυν δημοσιονομικών προοπτικών μέχρι το 2020. Είναι πρόημο να πούμε ότι υπάρχουν αυτά αποτελέσματα και ότι έχει υπάρξει και μια θετική εξέλιξη λόγω αυτού. Ε, έχουμε τα προγράμματα τα οποία έχουν λάβει σε χρηματοδότηση μέχρι τούδε το Ocean 2020 που σας ανέφερα ε, είναι κάτι το οποίο εξακολουθώ να επενώ γιατί έχουμε 42 επιχειρήσεις από την Ευρώπη και συμμετείχαν όλες σε κοινό πρόγραμμα και να υποβάλουν κοινό διαγωνισμό, κοινή προσφορά και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ξεκίνησε από την υποβολή της προσφοράς. Ε, θα σας δώσουμε τον κατάλογο των προγραμμάτων που είναι ακόμα στη διαδικασία υλοποίησης αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν Χάουαρτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε, για τις ε, παρατηρήσεις σας. Εγώ εκπροσωπώ μια περιφερεια του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει ε, υγιή ε, τομέα στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις ε, αεροπορικές εταιρείες και το αεροδιάστημα και φυσικά ε, συμμετέχουν στην παγκόσμια και στην ευρωπαϊκή ε, αλυσίδα αξιών και χαιρόμαστε ε, για τη συμμετοχή στην Ευρώπη, Αντιθέτω από κάποιου συναδέλφου. Έχω μία ερώτηση λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα, ε, το οποίο καλωσορίζω και καλωσορίζω και την πρόοδο που επετεύχθη και απορρίπτω και υπερβολικά σχόλια για απειλέ για την εθνική κυριαρχία και τα τι αυτά. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μα κάνει πιο ανθεκτικού, πιο αποτελεσματικού και εν τέλει και πιο ασφαλεί. Δύο ερωτήσει. Η μία αφορά την ευκαιρία ε, υποβιαμηχανικού όρου να μεγιστοποιήσουμε τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μεγιστοποιήσουμε και ε, το να παίρνουμε τα ε, διάφορα συστατικά στοιχεία και τα ανταλλακτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι το οποίο θα είναι προ όφελο Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και φυσικά και τη δική μου την περιφέρεια υπό την προπόθεση ότι θα παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσον διαβλέπετε απειλέ ε, από το Brexit. Το πρόγραμμα αυτό, ως έχει, θέλει να μεγιστοποιήσει τις πηγές και να ενισχύσει όλη την αλυσίδα αξιών. Το 70% του προγράμματος, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι αφιερωμένο σε μικρότερες επιχειρήσεις και καινοτόμες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ έχετε το ερώτημα της ε, αλυσίδας αξιών. Η όλη έννοια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας ε, και το πρώτο σκέλος το ερευνητικό και τις δημιουργίες ικανοτήτων στη συνέχεια. Ε, είμαι πολύ αισιόδοξη με τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί εμείς φοβόμασταν και φοβόμουν και εγώ προσωπικά στην αρχή, όταν ξεκίνησε το σκέλος της ε, έρευνας στην άμυνα, ότι δεν θα έχουμε προγράμματα, δεν θα αναπτυχθούν προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τόσους πολλούς εταίρους, οι οποίοι όπως σας είπα, ξεκινούν από την έρευνα και φτάνουν μέχρι την προμήθεια τελικά ε, των ικανοτήτων. Και προς ε, έκπληξή μας, η οποία ήταν και θετική, είχαμε πάρα πολλά προγράμματα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο από γεωπολιτική σκοπιά για να ενισχύσουμε την κυριαρχία μας και να έχουμε ε, καλύτερη ε, βοήθεια προς τους εταίρους μας να είμαστε ισχυρότεροι εταιρεία, αλλά και προς άλλες κατευθύνσεις. Σας παρακαλώ μην με ρωτάτε τώρα για τα αποτελέσματα του Brexit, τι να σας πω. Ναι, καταλαβαίνω πώς νιώθετε, ε, λέει ο κύριος Χόουερ. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα, δεν πριν από ένα χρόνο, πριν από έξι μήνες έλεγα ότι εάν υπάρχει γενική συμφωνία θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε σε κάθε κλάδο ξεχωριστά. Τώρα τι να σας πω. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου να μην απαντήσω και να μην σχολιάσω. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Άλλες ερωτήσεις? Επιτρέψτε μου να ρωτήσω κι εγώ λοιπόν, μετά από πέντε χρόνια ως Επίτροπος, ε, Πώς βλέπετε την προετοιμασία της Γενικής Διεύθυνσης ε, Βιομηχανίας Άμυνας και Διαστήματος. Θεωρείτε ότι διαθέτει πλέον κατάλληλες δεξιότητες για να μπορέσει να συστηθεί γρήγορα πώς βλέπετε τη διάρθρωσή της με τις άλλες ε, υπηρεσίες ε, στα άλλα θεσμικά όργανα που είναι αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και μία σύντομη ερώτηση γιατί αναφερθήκατε ακροθυγώς στην εισαγωγή σας σε θέματα διαστήματος και το ενδιαφέρον που έχετε γι' αυτό. Ίσως θα μπορούσατε να πείτε κάποια πράγματα για την εμπειρία σας ε, στα πέντε χρόνια σας ως Επίτροπος και να μας ε, δώσετε και κάποιες κατευθύνσεις για την επόμενη θητεία. Για τα θέματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα και στα οποία θα έπρεπε να επικεντρώσουμε και εμείς το ενδιαφέρον μας ε, στον τομέα της διαστημικής άμυνας. Ευχαριστώ. Για την πρώτη ερώτηση, Νομίζω ότι θα ζήσουμε συναρπαστικές στιγμές. Συζήτησα με τον διάδοχό μου και νομίζω ότι υπάρχει μια καλή βάση. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό από πολλού ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σίγουρα η γενική διάθεση αυτή θα χρειαστεί εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη, περισσότερους υπαλλήλους, διότι τα κονδύλια και ο τομέας που θα είναι τη αρμοδιότητάς τους θα είναι πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερος ο κλάδος από ό,τι γνώριζαν μέχρι τώρα. Όπως σας είπα, για πάνω από δύο χρόνια εμείς ε, προετοιμαζόμαστε για αυτή τη Γενική Διεύθυνση για να είναι κάτι ξεχωριστό. Ε, γιατί ήμουν απόλυτα βέβαιη ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή και νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε απαραίτητο, σίγουρα χρειαζόμαστε δυναμικό, χρειαζόμαστε γνώσεις, αλλά επιτρέψτε μου να το θέσω ως εξής. Ε, η γενικότερη νοοτροπία της άμυνας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν υπάρχει, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εμπλέκεται σε μια τέτοια διαδικασία διαχείρισης ενός τέτοιου προγράμματος. Επομένως, ε, είναι φυσικό και επόμενο ε, να πρέπει να αυξηθεί η εμπειρογνωμοσύνη. Όπως σας είπα υπάρχει πολύ καλό υλικό, αλλά είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρίως για το πεδίο του προγράμματος ε, που είναι ακόμα σε εξέλιξη και θα εξελιχθεί περισσότερο στα επόμενα δύο χρόνια. Όσον αφορά τις προτεραιότητες, βεβαίως, νομίζω ότι ε, δεν είμαι εγώ αυτή η οποία θα συμβουλέψω τι θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Νομίζω όμως ε, ότι και οι τρεις ή και οι τέσσερις αν θέλετε πλευρές, δηλαδή το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ίδιος ο κλάδος θα πρέπει να προσπαθήσουν να διατηρήσουν το ίδιο ανοιχτό, καλό και ειλικρινές ε, πνεύμα μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό ε, και είναι σημαντικό διότι πρέπει πραγματικά να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι θέλουν και οι άλλοι εταίροι. Δεν θέλω να του αποκαλώ άλλη πλευρά. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι θεώρησα ότι οι ερωτήσεις για επιχειρήσεις τρίτων χωρών ε, είναι περιτές, γιατί κάναμε πολλή προσπάθεια και επενδύσαμε πάρα πολύ ε, για να διευκρινίσουμε την ε, κατάσταση, αλλά και πάλι ανακύπτουν τέτοιες ερωτήσεις. Όλοι οι εταίροι λοιπόν θα πρέπει να έχουν ε, ετοιμότητα ε, και να απαντούν με ειλικρίνεια σε αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες ε, δεν είναι πάντα καλοπροαίρετες, αν θέλετε. Για, από τη δική μου την πλευρά η απάντηση είναι σαφής. Δεν πρόκειται για μέσο προστατευτικό, δεν κλείνουμε την αγορά μας, απλώς υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας σε θέματα ασφάλειας. Οι άλλοι πάνε πολύ παραπέρα, είναι πολύ πιο κοντά στις επιχειρήσεις μας. Ε, ε, αυτό που σχεδιάζουμε εμείς για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας. Ε, επομένως, σίγουρα θα έχουμε επιχειρήσει των χωρών. Ήθελα να προσθέσω μόνο διότι σιγά σιγά συσσωρευόντουσαν οι γνώσει μας για το πρόγραμμα αυτό. Και αν συμφωνείτε, πολύ ευχαριστώ να σας ε, καταρτήσω ένα κατάλογο ε, με τα προγράμματα, μια σύντομη ενημέρωση δηλαδή για το πώς ξεκίνησε το όλο θέμα, πώς εξελίχθηκε και με κάποιες ερωτήσεις και προτάσεις για το πώς μπορούμε να απαντήσουμε στις δύσκολες ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν από όλες τις πλευρές. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόταση, το εκτιμούμε ιδιαιτέρως και σίγουρα θα χρειαστούμε αυτές τις πληροφορίες για τη διαδρομή που ακολουθούσατε, αλλά φυσικά και με την σφραγίδα της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε για τα θέματα τα οποία κρυμούν ακόμα και διότι τρόπον την να κάνατε περισσότερα από το να ανοίξετε απλώς το δρόμο ε, και δείξατε και την κατεύθυνση στη διάρκεια της δικής σας της θητείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματικά ε, χρειαζόμαστε και την ε, παρακαταθήκη σας τα έλεγα ως Επίτροπος αλλά ναι ναι, αυτό ήταν πολύ σημαντικό σκέλος του χαρτοφυλακίου μου. Εκτιμώ φυσικά τα όσα έγιναν, όχι μόνο από μένα, από τους υπαλλήλου μου, από τις υπηρεσίες μου, από το Συμβούλιο, από το Κοινοβούλιο και από αυτή την Επιτροπή στην προηγούμενη θητεία. Και φυσικά βασίζομαι και στην υποστήριξή σας για το μέλλον αλλά και για το διαδοχό μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της σταδιοδρομίας σας.

Συνάδελφοι, η Επιτροπή Αμυντικών Θεμάτων καλωσορίζει θερμά τον κύριο Πάβελ Χερτσίνσκι, Γενικό Διευθυντή της ΠΕΣΚΟ, για τις αστικές της αποστολές, που είναι και οι πιο συχνές επιχειρήσεις ε, που γίνονται σήμερα υπό την ΠΕΣΚΟ και που είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και συνεισφέρει στην ειρήνη και στην ασφάλεια. Την PSDC. Υποστηρίζοντας ε, τους, ε, τις χώρες εταίρους ώστε να υποστηρίζουμε την ειρήνη και την ασφάλεια και στο δικό τους έδαφος συνεισφέροντας και στη δική μας ειρήνη και ασφάλεια είχαμε ένα νέο σύμφωνο αστικής συνεργασίας στα πλαίσια της ε, αμυντικής ε, συνεργασίας και συνεργασίας θέμα της ασφαλείας, της PSDC, ώστε να υποστηρίξουμε την, τόση σχετισμό μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και να έχουμε μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των αστικών αποστολών και Τη συνεργασία με τα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών. Χρειαζόμαστε λοιπόν την απαραίτητη οργάνωση για την καλύτερη διαχείριση των αποστολών. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία συνεισφέρουν στην επιτυχία του συμφώνου αυτού. Πέρα από τις ε, παραδοσιακές τους εντολές ε, για τις ε, αστυνομικές δυνάμεις, τις αστικές επιχειρήσεις και τα δικαστικά θέματα, έχει και νέες εντολές σχετικά με τα θέματα μετανάστευσης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της τρομοκρατίας ε, και της ριζοσπαστικοποίησης. Όπως και της ασφάλειας της θάλασσης, ε, την πρόληψη στον ε, βίαιο εξτρεμισμό και στην προστασία του πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης διαθέτουν τις απαραίτητες επιχειρησιακές αυτές δυνατότητες που χρειάζονται ώστε να προχωρούμε σε, σε αποστολές 200 ατόμων εντός 30 ημερών μετά από μια απόφαση του Συμβουλίου με τον απαραίτητο εξοπλισμό που παρέχεται σε στρατηγικό επίπεδο. Επεξεργαστήκαμε ε, ένα κοινό σχέδιο δράσης για την PSDC που προβλέπει 74 δράσεις για τις 22 εντολές που συμπεριλαμβάνονται στο σύμφωνο αυτό, ώστε να έχουμε μια πλήρη εφαρμογή και στους ερχόμενους μήνες τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγκρίνουν σχέδια δράσης εθνικά που θα είναι φιλόδοξα και που θα έχουν και τους απαραίτητους πόρους χρηματοδότησης που θα ανταποκρίνεται στο επίπεδο φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κύριε Τσίνσκι, θα θέλαμε να μα ενημερώσετε για το πώ έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή με την εφαρμογή του συμφώνου συνεργασία, ποιε είναι οι βασικέ δράσει που συμπεριλαμβάνονται και σε ποιο επίπεδο, μάλλον τι επίπεδο δέσμευση περιμένετε ή προσδοκάτε από τα κράτη-μέλη. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων που σα έχουν ανατεθεί ιδιαίτερα στα θέματα άτυπης μετανάστευσης, διαχείριση των συνόρων και όλα τα προηγούμενα που ανέφερα, ποιες συγκεκριμένε δράσεις προβλέπετε για να έχουμε καλύτερη, πιο αποτελεσματική συνέργεια με τους φορείς ε, των θεμάτων δικαιοσύνης και εσωτερικών των κρατών μελών, ώστε να επιτύχετε τους στόχους που έχουν τεθεί μαζί με τους παραδοσιακούς στόχους ε, της αστικής, ε, δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Το θεματολόγιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Θα μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε αν αν έχουν διατεθεί απαραίτητα μέσα, επαρκή μέσα, ώστε να επιτεθούν. αυτοί οι στόχοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι τιμή για μένα που μπορώ και σας μιλώ σήμερα εδώ στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ονομάζομαι Πάβελ Χερτσίνσκι. Μόλις ορίστηκα Γενικός Διευθυντής του CSDP και τη διαχείρισης κρίσεως ε, της Υπηρεσίας εξωτερικών Δράσεων. Έχω και την συνάδελφο Γιάννεκ Μπρόβερ, εδώ δίπλα μου, η οποία είναι εμπειρογνώμων σε αστικά θέματα συνεργασίας. Ε, έχει εργαστεί με διάφορες αρμοδιότητες στα θέματα αυτά εδώ και αρκετό καιρό. Σας ευχαριστώ θερμά για την εισαγωγή σας. Έχετε θέσει το σωστό, το απολύτως σωστό πλαίσιο της συζήτησης. Οι αστικές στοιχείες του CSDP είναι μια προστιθέμενη αξία για τον διεθνή ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα ασφάλειας και ειρήνης. Επί τη βάση των 16 ετών εμπειρίας τα αιστικά αυτά προγράμματα συνεργασίας πρέπει να ενισχυθούν, αυτό αισθανόμαστε όλοι, δεδομένος, δεδομένων με των μεταμορφώσεων του στρατηγικού γεωπολιτικού περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ανάδυση διαφόρων ζωνών ε, συγκρούσεων γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασυνοριακών απειλών και κινδύνων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα ποιοτικό και ποσοτικό άλμα στα αστικά θέματα του CSDP ώστε να ενισχύσουμε το ρόλο της Ένωσης ως ε, διεθνή παίκτη στα θέματα διαχείρισης κινδύνου σε αστικό επίπεδο. Είναι ένα θεμελιώδες ε, στοιχείο στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με άλλα μέσα, ολοκληρωμένα και όλα αυτά προς την κατεύθυνση της ε, παγκόσμιας στρατηγικής για τα θέματα ασφάλειας και ειρήνης, που είναι το γενικό μας σύνθημα. Η συνολική στρατηγική αυτή είναι μια ομπρέλα και πηξίδα των δράσεών μας, ώστε να επενδύουμε περισσότερο σε δράσεις αστικού, αστικής συνεργασίας. Το Συμβούλιο το περασμένο Δεκέμβριο υπέβαλε αυτό το σύμφωνο με δεσμεύσεις για την ενίσχυση της αστικής συνιστώσας του CSTP. Συμπεριλαμβάνει 22 πολιτικές δεσμεύσεις του Συμβουλίου και των κρατών μελών ε, για την ανάληψη ενός αριθμού δράσεων με βασικό στόχο οι αστικές αυτές επιχειρήσεις να είναι πιο αποτελεσματικές με τη δέσμευση των κρατών μελών ανάπτυξης του απαραίτητου δυναμικού, διαχείρισης, καλύτερης διαχείρισης του προσωπικού και πιο ευέλικτης ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε διάφορες κρίσεις συνολικά και από κοινού με άλλα ευρωπαϊκά μέσα υπό την ολοκληρωμένη αυτή προσέγγιση αντιμετώπισης κρίσεων σε στενή συνεργασία με άλλους φορείς τζάι ε, εσωτερικών θεμάτων και θεμάτων δικαιοσύνης αναφερθήκατε στους 2.000 στρατιωτικό προσωπικό έχουμε πράγματι Στρατιωτικού στις επιχειρήσεις μας, στι αποστολέ μα, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ένα στρατιωτικό υπόβαθρο η εμπειρία, αλλά προέρχονται από τις αστυνομικές δυνάμεις, από τις δικαστικές δυνάμεις, από τη συνοριοφυλακή, από διάφορα σώματα. Για να υλοποιήσουμε λοιπόν και να εφαρμόσουμε το σύμφωνο αυτό, η ΕΔΕ και η Επιτροπή εργάζονται μέσω κοινού σχεδίου δράσεως, για να υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη για τους στόχους του συμφώνου. Η πρώτη ετήσια έκθεση δυναμικού για τις αστικές επιχειρήσεις θα μας δώσει μια συνολική εικόνα των δυνατοτήτων που έχουμε και θα ενημερώσει τα κράτη-μέλη για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Επιπροσθέτως, συνεχίζεται η δουλειά ώστε να ενισχύσουμε την συνεργασία με τους φορείς ε, της εσωτερικής ασφάλειας και τις ενίσχυση του συσχετισμού μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής. Έχουμε λοιπόν κάποια ούτως αποκαλούμενα μίνι σκεπτικά που σχετίζονται με την άτιμη μετανάστευση, τις υβριδικές απειλές, ε, την, ε, ε, το κίνδυνο στον κυβερνοχώρο, τη διαχείριση των συνόρων, τη διαχείριση των θαλασσών, την ασφάλεια των θαλασσών και την ανάγκη της προστασίας της πολιτικής κληρονομιάς. Ε, μια πρόκληση εδώ <clears throat> είναι η ομαδοποίηση των φορέων που έχουμε στη διαθέσή μας και μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας, όπως η Frontex, που προβλέπει αποζημίωση για την απόσπαση προσωπικού από τα κράτη-μέλη για τέτοια προγράμματα ή αποστολές, ε, μοίρασμα των πόρων, κοινό αποθεματικό πόρων δηλαδή, και αποτελεσματικές και πλήρες συνεργα... Ε, συμφωνίες μοιραζόμαστε δηλαδή τους πόρους με τα κράτη-μέλη και στην ουσία, για να το πούμε ειλικρινά, ανταγωνιζόμαστε. Ίσως να μην είναι πολιτικά ορθή η ορολογία αυτή, αλλά έτσι περίπου έχουν τα πράγματα. Χρειαζόμαστε ευέλικτε αποστολέ που να προσαρμοστούν σε κάθε επίπεδο στόχου, ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματικά, οικονομικά πιο αποτελεσματικέ και επιχειρησιακά πιο αποτελεσματικέ αποστολέ, ώστε να έχουμε καλύτερη διαχείριση των προσωπικών λογισμικού, ανθρωπίνων πόρων, επιλογής έργων. Ο ρόλος των κρατών μελών, και εδώ απαντώ στην ερώτησή σας, είναι κρίσιμος. Έχουμε αποσπασμένους εμπειρογνώμονες στην κοινή πολιτική ε, ασφάλειας και ειρήνης, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια μόνο 10 κράτη-μέλη έχουν αποσπάσει περί το 70% των εμπειρογνωμόνων αυτών. Αριθμό που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αποστολών. Ε, το σύμφωνο έχει δημιουργήσει φορεί συνεργασία στα κράτη-μέλη, αν θέλετε για να πούμε έτσι, η επικοινωνία, αυτό είναι ελπιδοφόρο, θετικό σημάδι. Ένα αριθμό κρατών μελών να αναπτύσσουν περαιτέρω τα δικά του συστήματα για να ανταποκρίνονται καλύτερα τις ανάγκες, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο, τους χρηματοδοτικού τους ε, πόρους και βεβαίως την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Η επιφάνεια της εθνικής ε, συνεισφοράς ε, με προσωπικά αποσπασμένο και στρατηγική επικοινωνία θα μπορούσε να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο την τάση αυτή. Τα κράτη-μέλη στο πρώτο συνέδριο της ετήσιας έκθεσης που θα γίνει τον Νοέμβριο φέτος θα ανταλλάξουν απόψεις και πρέπει να διατηρήσουμε την όθηση αυτή, την τάση αυτή προς το 2023 όπως έχουμε συμφωνήσει με τα κράτη-μέλη. Προτού ολοκληρώσω θα πω σύντομα ε, δύο λόγια για τα του μέλλοντος. Στο Σύμφωνο Αστικής Συνεργασίας το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη συνεφώνησαν να έχουν μια πρώτη συνάντηση για τα αστικά τα αυτά προγράμματα στο δεύτερο εξάμεινο του 2019, για να σημειώσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί και να γίνει μια προτεραιοποίηση προς το μέλλον. Αυτή η πρώτη, το πρώτο ετήσιο συνέδριο θα γίνει 14 Νοεμβρίου. Θα σημειώσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί, τη δουλειά που έχει γίνει και εδώ στην έδρα αλλά και στις επιμέρους έδρες των κρατών μελών και θα διαμορφώσουμε ένα φύλλο πορείας για τα επόμενα χρόνια ώστε τα κράτη-μέλη και οι υπηρεσίες της Επιτροπής να δρουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα εντό στα πλαίσια του συμφώνου. Με ενδιαφέρον είμαι στη διάθεσή σα για το υπόλοιπο τη συζήτηση. E. Ο κύριο Ντανζάν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Χαίρομαι που έγινε πλήρης αναθεώρηση των πολιτικών αποστολών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό Θεωρώ ότι αυτή που επιτροπή όταν ε, ασχολήθηκε με θέματα τέτοιων πολιτικών αποστολών έλαβε υπόψη τις, ε, τις αποστολές που είχαν γίνει σε όλες τις χώρες ε, που είχαμε τέτοιες αποστολές και πολλές φορές είχαμε ακολουθήσει πολύ εύστοχα επιχειρήματα. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία πράγματα. Το ένα είναι αμυγός πολιτικό, το οποίο δεν το συζητάμε τόσο ένα από τα προβλήματα αυτών των αποστολών είναι ότι η εκφύσεως είναι πολύ συχνά, αυτό είναι, δεν είναι δική σα ευθύνη βέβαια, είναι των κρατών μελών, πολύ συχνά θεωρούνται ω αποστολέ λόγω προβλήματο. Δηλαδή έχουμε μια κρίση κάπου, ξεκινάει μια στρατιωτική αποστολή, μάλλον το να γίνει στρατιωτική αποστολή είναι πολύ σύνθετο και έχει και άλλε προεκτάσει πέραν τη κρίση. και επομένω είναι η ίστατη λύση και τόσο το καλύτερο, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και απόντες από την κρίση. Ε, τα παραδοσιακά διπλωματικά μέσα, οι αντιπροσωπείε μα η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν επαρκούν. Επομένως, χρειάζεται ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσης, πολιτική αποστολή. Και εκεί δεν τίθεται τόσο πολύ το ερώτημα του κατά πόσον ε, είναι τέλεια σχεδιασμένη η αποστολή ε, ε, υπάρχει απλώ πολύ συχνά η πρόκληση το να πάμε να στήσουμε την ευρωπαϊκή στιμία και να πούμε ότι είμαστε παρόντες εκεί. Ε, και κάπου ε, αποφασίζοντας μια πολιτική αποστολή ε, νύπτουν τα σχήρα του οι υπόλοιποι και θεωρούν ότι έληξε το πρόβλημα. Εμείς ε, πιστεύουμε ότι ίσως θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα και να είναι ε, αποστολές οι οποίες γίνονται για να επιλύσουν το πρόβλημα, όχι για να πούμε ότι είμαστε εκεί. Ε, και υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό στα συμπεράσματα τα οποία εγκρίθηκαν και το υπενθυμίσατε κι εσείς νομίζω το να υπάρχει μία ε, κλιμακωτή και ανά την περίπτωση εντολή. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο εξαλίσσεται η αποστολή να προσαρμόζεται συνέχεια και η δυσκολία ακριβώς αναπροσαρμογής των ε, αποστολών αυτών μπορεί να σημαίνει και ορισμένες φορές ότι θα πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι άγνωστο, ας πούμε, ότι εγώ πολύ συχνά είχα πάρα πολλές ε, επικρίσεις για τις αποστελές μας ε, στο Αφγανιστάν. Εγώ αμφισβητούσα την ύπαρξή τους, αλλά ξεκίνησε κάτι όπως σε όλες τις οργανώσεις. Υπήρχαν και πολιτικά θέματα από κάποιες χώρες οι οποίες μπλόκαραν κάποια πράγματα και χρόνο, ενέργεια και αξιοπιστία για, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον των εταίρων μα. Και νομίζω ότι ε, έχουν γίνει κάποια βήματα προ τη σωστή κατεύθυνση, έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα προ τη σωστή κατεύθυνση. Δύο ακόμα παρατηρήσει πολύ σύντομα. Όσον αφορά το κόστο δεν είναι καθόλου πολιτικά, είναι πολύ συγκεκριμένο και είναι και εμπειρικό σε σχέση με την εμπειρία που είχα. Εγώ επισκέφθηκα όλε τι πολιτικέ αποστολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και ακόμα και πριν γίνω Ευρωβουλευτής ε, είχα υπηρετήσει σε κάποιες από αυτές και εργάστηκα σε κάποιες από αυτές. Και αυτό το οποίο ε, με εξέπλητε κάθε φορά ήταν το ίδιο πρόβλημα. Συγκεκριμένο πρόβλημα τοπικής διαχείρισης των χρημάτων, των ανθρωπίνων πόρων, του εξοπλισμού ε, με ε, κάποιες περιπτώσεις στις οποίες ε, τρελαινόταν ο υπεύθυνο για να διαχειριστεί την κατάσταση στη χώρα υποδοχής της αποστολής. Έχουμε αναρρύθμιτα παραδείγματα και χρημάτων και ενέργειας που χάθηκαν και σπαταλήθηκαν ε, για θέματα ε, απλώ διαδικασία. Πρέπει να υπάρχουν διαδικασίε, πρέπει να υπάρχει έλεγχο γιατί μπορεί να υπάρξουν καταχρήσεις, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να είμαστε πολύ ρεαλιστέ και πολύ ελαστικοί στη διαχείριση για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε όλε τι συνθήκε που θα αντιμετωπίσει ο τόπου. Διότι εκφύσεως είναι αποστολέ για διαχείριση κρίσεων που και δεν έχουμε αντιμετωπίσει με την ίδια κατάσταση που έχουμε και στι Βρυξέλλε. Εδώ και 20 χρόνια όπου και αν πάμε το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Ε, αγορά, για παράδειγμα, χρηματοκιβωτίου στη Σομαλία, αγορά υλικού ε, εξοπλισμού επικοινωνίας στο Μάλι. Ε, όλες οι αποστολές αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν και χάνουν πάρα πολύ ε, ενέργεια και χρόνο εκεί. Και ένα τρίτο σημείο και πάλι τεχνικής φύσεως, η παρακολούθηση των αποστολών αυτών, η συνέχεια. Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι. Εγώ πάντα ε, καλωσορίζω αυτόν τον επαγγελματισμό. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι στέλνονται σε αυτές τις αποστολές. Η χώρα υποδοχή, αν θέλετε, δυστυχώς ε, γίνεται μια εξαιρετική κατάρτιση, δίνονται κάποιες εξαιρετικές στρατηγικές ε, ε, συμβουλές, αλλά είναι μια φορά και μόνο και δεν υπάρχει καμία παρακολούθηση. Υπάρχει για παράδειγμα το παράδειγμα στο, στο Νίγηρα. Οι αστυνομικοί της Νιγηρίας τότε μας έλεγαν ότι από όλες τις εκπαιδεύσεις που μας κάνατε η εκπαίδευση της ε, αστυνομίας σε θέματα ε, κλιματικότητας ε, και σήμανσης ήταν η πιο σημαντική γιατί έγινε χάρη στα εργαστήρια, σε υπολογιστές, τα οποία όμως δεν μας στείλανε μετά. Μας εκπαιδεύσανε για αυτά και δεν μας τα στείλανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν κάνει αυτό το εξαιρετικό πράγμα και τους εκπαιδεύει και μετά δεν υπάρχει καμία συνέχεια σε μια άλλη χώρα της Αφρικής, σε μια αντίστοιχη πολιτική αποστολή, είδαμε εκπαίδευση, η οποία έγινε και μετά εστάλει κινέζικος και τουρκικός εξοπλισμός δωρεάν από αυτούς τους γενναιόδωρους δωρητές που δεν μπορέσαμε εμείς, ε, ε, εκεί που δεν μπορέσαμε εμείς να δώσουμε βοήθεια. Υπάρχουν κάποια πράγματα οποία γνωρίζετε εσείς πάρα πολύ καλά, είναι πολύ συγκεκριμένα, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Ε, θα, θα έχουμε μεγαλύτερα αποτελεσματικότητα στις αποστολές μας αν τα λύσουμε αυτά τα πράγματα και μεγαλύτερη εξοπιστία σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίξερ. Uh, um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πολύ καλή παρουσίαση. Δύο ερωτήσεις έχω. Από ό,τι είπατε, το σύμφωνο προέκυψε από τη συνειδητοποίηση ότι τα κράτη-μέλη σιγά σιγά άρχισαν να φθήνουν ως προς τη συμμετοχή τους σε αυτές τις πολιτικές αποστολές και τώρα ε, χάρη στο σύμφωνο είχαμε μια νέα ε, όθηση. Και καλό είναι να καθορίσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας ε, για τη συμβολή μας σε αυτές τις πολιτικές αποστολές. Πριν από πολλά χρόνια, θυμάμαι, στα βάθη του άλλου φάσματος, στη στρατιωτική πλευρά, όταν το ΝΑΤΟ είχε την έννοια των NRF, στοιχεία τα οποία υποτίθεται θα μπορούσαν να σταλούν εντός πέντε ημερών. Πρόκειται για τεράστια φιλοδοξία και Κάποιο είπε κάποια στιγμή ότι το να έχουμε δυνάμει σε έτοιμο πόλεμε εντό πέντε ημερών είναι πάρα πολύ δαπανερό και ακόμα και αν έχεις τις ε, διαδικασίες που σου επιτρέπουν να λάβεις την πολιτική απόφαση, ε, χρειάζονται τουλάχιστον πέντε μέρε, αλλά πολύ περισσότερες από τις πέντε μέρε. Φαντάζομαι ότι αυτοί οι εμπειρογνώμονες πολίτες ε, που μπορούμε να στέλνουμε κοιμούνται έτοιμοι, για να φύγουν σε κάποια αποστολή ανά πάσα στιγμή. Θα ήθελα να ξέρω τι φιλοδοξίες έχουμε ως, ως προς τις δυνατότητες μας και την ικανότητα να λάβουμε τις αποφάσεις που χρειάζονται για να ε, ε, ξεκινήσουμε αυτές τις αποστολές. Η δεύτερη ερώτηση ε, προκύπτει από την προηγούμενη ερώτηση του συναδέλφου Ντανζά. Πολύ συχνά Προσπαθούμε να βγάλουμε του αυτού μα έξω από αυτέ τι ε, σειράξει, συγκρούσει. θέλουμε κι εμεί και δεν θέλει ο φορολογόμενο να έχει ανοιχτέ δεσμεύσει. Θέλουμε να τελειώσει κάποια στιγμή η αποστολή και να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να βγούμε εμεί στην άκρη. Και φυσικά αυτό είναι προφανέ με στρατιωτικέ επιχειρήσει, αλλά όταν είναι πολιτική αποστολή μπορεί να είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Παραδείγματο χάρη, αποστολέ ε, για εκπαίδευση. Ε, στην ε, λαϊκή ε, Δημοκρατία της Αφρικής, για παράδειγμα, μια ε, αποστολή εκπαίδευσης που κάναμε, και ξέρουμε ότι εκεί υπήρχε ευγενή στόχος να δημιουργήσουμε ικανότητες για τους αυτόχθονες στην περιοχή και κάποια στιγμή φάνηκε ότι τα ωφέλη τα εκμεταλλεύτηκε κάποιος εξωτερικός παίκτη, ο οποίος είναι πολύ, είχε πολύ πιο χαμηλότερες προσδοκίες σε σχέση με εμάς η γεωστρατηγική του στόχη ήταν τελείως διαφορετική από τους δικούς μας. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς ε, να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα διακινδυνεύσουμε να χάσουμε όλη αυτή την προστιθέμενη αξία που δημιουργήθηκε μετά την αποστολή, αμέσως μετά την αποστολή, ε, με το πέρας δηλαδή της αποστολής. Ο κύριος Οστρεβίτσιος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Αναφερθήκατε σε ποια κράτη-μέλη έχουν συμβάλει κατά πόσο. Είπατε 10 κράτη-μέλη το 75% και τα άλλα 18 δηλαδή το 25%. γιατι τόσο τόσα πολλά κράτη-μέλη δεν συμμετέχουν πιο ενεργά. Και οικονομικά δεν έχουν πόρους δηλαδή. Δεν έχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες και προσωπικό, πολιτικές αμφιβολίες για ιστορικούς λόγους κάποιων κρατών μελών. Δεν θέλουν να εμπλακούν σε κάποιες ε, περιοχές δηλαδή. Λέτε ότι τα κράτη-μέλη βεβαίως πρέπει να σας δώσουν τις δυνατότητες για να αντιμετωπίσετε κρίσεις. Υπάρχει κάποια κοινή στρατηγική. Κάποια απόπειρα να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν αυτές τις δυνατότητε. Ή κυρίως ε, επαφείται σε κάθε κράτος μέλος, βέβαια καταλαβαίνω, επαφείται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει. Αλλά κάνουμε τίποτα ως ένωση για να έχουμε τις δυνατότητες στην κατάλληλη στιγμή και του κατάλληλου επίπεδου. Ο κύριος Βατσικόφσκι από το ECR. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χαρτσίνσκι για τη σύντομη παρουσίασή σας. Μα γνωριζόμαστε. Ξέρετε, λοιπόν, ε, εφόσον γνωριζόμαστε, καταλαβαίνετε ότι οι ερωτήσει μου θα είναι προκλητικές και σταράτες. Έχετε αυτούς τους 2.000 στρατιωτικούς και πολιτικούς ε, εμπειρογνώμονες. Τι έχετε επιτύχει με όλους αυτούς. Αυτός ο στρατός εμπειρογνωμόνων ποιες κρίσεις έχει επιλύσει τα τελευταία χρόνια. Ποιους προστατεύσατε με το μηχανισμό αυτό. Τι αποτρέψατε. Κυβερνοεπιθέσεις για παράδειγμα ή άλλου τύπου επιθέσεις. Ε, γιατί έχω την εντύπωση ότι συζητάμε κάτι που είναι σε επίπεδο πολύ θεωρητικό. Είπατε ότι έγιναν αποστολές, είπατε ότι έχετε εμπειρογνώμονες. Ε, κάτι κάνουν. Ε, τι έχουν επιτύχει. Τι επέτυχαν οι αποστολές στις οποίες αναφερθήκατε. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω μία ερώτηση κι εγώ για τις επιπτώσεις του Brexit στις πολιτικές αυτές αποστολές CSDP, δηλαδή κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τι επιπτώσεις θεωρείτε ότι θα έχει το Brexit. Τι προβλέψεις έχετε κάνει για τις αποστολές σας. Ευχαριστώ πολύ. Μα θαυμάσεις ερωτήσεις. πολιτικές στην ουσία τους. Λοιπόν, θα απαντήσω. Αλλά καταρχάς μια γενική παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις ε, ελάχιστες διεθνείς οργανώσεις που έχει τη δυνατότητα, έχει το κατάλληλο εξοπλισμό για να δρά εκτός της επικράτειάς της. Εφόσον βεβαίως υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση των κρατών μελών. Φυσικά υπάρχουν και τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή είναι το, ο, ο κυριότερος παρεμβαίνων μέσω των ειρνευτικών αποστολών. Αλλά αν εξαιρέσουν τα Ηνωμένα Έθνη, μετά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και η Αφρική Ένωση που είναι ακόμη στα σπάργανα οι απόπειρές της είναι ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν ειρνευτικές αποστολές. Και κανείς άλλος. Νομίζω ότι το να έχουμε στο οπλοστάσιό μας και στρατιωτικές και μη στρατιωτικές αποστολές, το δυνατότητα δηλαδή να κάνουμε τις αποστολές, είναι θεμελιώδες. Μπορούμε να συζητήσουμε ποια είναι η επίπτωση επιτόπου. θα κάνουμε σοβαρά όλα αυτά. Μήπως είναι όλα αυτά προπέτασμα καπνού. Είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Καλά, αυτό είναι θέμα εκτίμησης του καθενός. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια κάναμε πάνω από 30 διαφορετικές αποστολές. Αυτή τη στιγμή είναι εν εξελίξη 16. Περισσότερες πολιτικές. Και προσπαθούμε να έχουμε επιπτώσεις επιτόπου. Σε τρεις υπήρους ε, ενεργούμε. Καμιά φορά είναι μόνο σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις ανάγκες. Αλλά στην τελευταία ανάλυση αυτό είναι θέμα βούλης των κρατών μελών. Εξαρτώμεθα από τα κράτη-μέλη. Όπου υπάρχει βούληση, όπου υπάρχει φιλοδοξία, όπου υπάρχει ετοιμότητα να συμβάλλουν, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Παραλαμβάνω, εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Πάντα βέβαια στέλνουμε μέσω των αποστολών αυτών ένα πολιτικό μήνυμα. Για παράδειγμα, Ουκρανία. Αποφασίσαμε να υπάρξει μια τέτοια αποστολή στην Ουκρανία μετά την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας. και μετά τη σύραξη στην περιοχή Ντόν Να βοηθήσουμε, αποφασίσαμε την Ουκρανία να αναπτύξει μη στρατιωτικές δομές γιατί όλοι ξέρουμε τι υφίσταται η Ουκρανία, τι προβλήματα υπάρχουν, ε, προβλήματα με το κράτος δικαίου, θέματα διαφθοράς. Γι' αυτό πηγαίνουμε και σε πολλά μέρη στην Αφρική και τα κράτη-μέλη συζητούν για το ενδεχόμενο να πάει μια πολιτική αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Είναι απελπιστική κατάσταση σε αυτή τη χώρα και υπάρχουν και άλλοι εκεί. Ίσως ε, με περισσότερους πόρους και οικονομικούς πόρους. Αλλά βεβαίως εμείς ε, θέλουμε να κάνουμε πολλά εμείς ως ε, θεσμοί της Ένωσης. Αλλά δεν έχουμε δικούς μας πόρους, δεν έχουμε δικό μας προσωπικό. Τα κράτη-μέλη πρέπει να το παράσχουν. Να τους παράσχουν και τους πόρους και το προσωπικό. Για τα τεχνικά και διαδικαστικά προβλήματα που έχουμε στις ε, αποστολές μας. Υπάρχει μια ειδική μονάδα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι η λεγόμενη δυνατότητα προγραμματισμού και σχεδιασμού αποστολών επικεφαλής ένας Ιταλός στρατηγός, ο Βιντσέντσο Κόπολα. Και επειδή υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για τα, αυτά τα συγκεκριμένα πρακτικά θέματα, θα σας πρότεινα να τον προσκαλέσετε για να σας ενημερώσει. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία προσπαθεί να βελτιώσει τις διαδικασίες, να είναι πιο ορθολογική η διεξαγωγή των αποστολών, να υπάρχουν ε, διαδικασίες που να ισχύουν για όλες τις ε, πολιτικές αποστολές και για να γίνει βέλτιστη χρήση των ε, υφισταμένων πόρων. Κάποιες αποστολές βέβαια πηγαίνουν, κάνουν τη δουλειά τους και μετά αποχωρούν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα μετά που έχουν αφήσει. Αυτή, αυτό το μέλημα είναι αυτό που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μέσω της λεγόμενης ολοκληρωμένης προσέγγισης. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Όταν υπάρχει κάπου μια κρίση θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με όλες τις δυνατότητες που έχουμε. Που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας όχι μόνο η υπηρεσία εξωτερική δράση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα. Προσπάθεια μεσολάβηση, ε, αποτροπή σειράξεων, αποστολή δική μα, ε, μέτρα ειρήνευση, ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια και εμπόριο. Έτσι προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα. Βέβαια, άλλο να το λες, άλλο να το κάνεις. Συμφωνώ. Αλλά αυτό είναι το υπόδειγμα το οποίο θα θέλαμε να εφαρμόσουμε. Έγινε μια σύγκριση με το λεγόμενο NRF και αυτή η ετοιμότητα πέντε ημερών. Όχι, όχι, είμαστε σε εντελώ άλλο πλανήτη. Συγχωρείτε που τα λέω απερίφραστα. Πρώτα απ' όλα, χρειαζόμαστε να συμφωνήσουν 28 κράτη-μέλη για να ξεκινήσει μια αποστολή. Κάποιο κράτος μέλος, συνήθως ή μια ομάδα κρατών μελών, Αναλαμβάνω την πρωτοβουλία για κάποιους λόγους, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, μετά γίνονται συζητήσεις σε ομάδες εργασίας και μετά πρέπει να ληφθεί μία ομόφωνη απόφαση για να ξεκινήσει μία αποστολή. Αυτό παίρνει χρόνο. Μπορούμε να παρεύουμε πολύ σύντομα, αλλά όχι σε πέντε μέρες, είναι άλλο επίπεδο. Και λυπάμαι γι' αυτό. Θαυμάσιο θα ήταν να μπορούσαμε να αναπτύξουμε μία αποστολή πολύ σύντομα. Αλλά ξέρετε, αυτές οι συζητήσεις παίρνουν εβδομάδες ή και μήνες. Και χρειάζεται ομοφωνία. Τι προβλήματα υπάρχουν με τα κράτη-μέλη και γιατί κάποια κράτη-μέλη συμβάλλουν περισσότερο από άλλα. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλα τα κράτη-μέλη είναι η διαθεσιμότητα κατάλληλου προσωπικού. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ένα άλλο. Τα περισσότερα κράτη-μέλη θέλουν να στείλουν προσωπικό. Αλλά όταν επιστρέφει αυτό το προσωπικό, μετά υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρουν τι να τους κάνουν, σε ποια θέση να τους ε, βάλουν. Στην περίπτωση των στρατιωτικών αποστολών είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Γιατί αν είσαι τμήμα μιας αποστολής, αυτό είναι τμήμα της σταδιοδρομίας ε, ενός στρατιωτικού. Αλλά τώρα για δημοσίους υπαλλήλους μη στρατιωτικούς όσοι συμμετέχουν σε αποστολέ, στην ουσία διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο ότι θα αποκοπούν από τις ε, διοικήσει των οποίων είναι μέλη. Θα συμμετάσχουν σε μια τέτοια αποστολή, θα γυρίσουν, μετά δεν έχουν θέση και πρέπει να ψάξουν για μια θέση. Αυτό είναι μια δυναμία, Την εντοπίσαμε με τα κράτη-μέλη και προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε μέσω της ανταλλαγής βελτίστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών. Και ένα κράτος μέλος εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει ένα κέντρο αριστείας για να γίνει μια συζήτηση, μια ανταλλαγή απόψεων, διαδικασιών που εφαρμόζονται σε διάφορα κράτη-μέλη. Κατόπιν. Για παράδειγμα. Πάμε κάπου, κάνουμε μια εκπαίδευση και μετά φεύγουμε. Και μετά τι γίνεται. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Έχουμε μια νέα πρωτοβουλία γι' αυτό. Την οποία ε, ξεκίνησε η αντιπρόεδρος Μογκερίνη που λέγεται Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση για την ε, Ειρήνη. Είναι σε επίπεδο συζήτησης μεταξύ κρατών μελών, δεν έχει εγκριθεί ακόμη, αλλά είναι η πρότασή μας για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και προτείνουμε 10,5 δισεκατομμύρια για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ένας από τους πυλώνες του, πυλώνες της αυτής της διευκόλυνσης, θα είναι η Ένωση να μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται μετά. Όχι απλώς να χορηγεί, ας πούμε, εκπαίδευση. Αλλά μετά να στέλνει και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ επίμαχο βεβαίω, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει αυτέ τι συζητήσει. Συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και φωνικών όπλων. Οι συζητήσει ε, συνεχίζουν μεταξύ 100 μελών, αλλά αν είμαστε σοβαροί για το ότι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο να παρέχει ασφάλεια, πρέπει να γίνει και αυτό. Πρέπει να συζητήσουμε αν τα 10,5 δις ε, επαρκούν, ή είναι υπερβολικά, ή είναι λίγα. Αλλά αν ε, θέλουμε σοβαρά να επιτύχουμε αυτό το στόχο, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας θα είναι εκτός προπολογισμού αυτό το ποσό. Κάτι που κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση σημαίνει επιπλέον πόροι να διατεθούν από τα κράτη-μέλη. Α, είστε ο πρώην προϊστάμενός μου. Σε ευχαριστώ για τις ε, θαυμάσεις ερωτήσεις σας. Τι έχουμε επιτύχει. Κάθε αποστολή είναι διαφορετική. Και μπορούμε να συζητήσουμε Εάν όντως, όντως αλλάζουμε τα πράγματα επί τόπου, έχουν επιπτώσεις, είναι μια τρύπα στο νερό. Ας πούμε για παράδειγμα για την αποστολή μας στη Γεωργία. Χθες ακριβώς με επισκέφθηκε ο επικεφαλής της αποστολής. Ο τρέχον επικεφαλής. Μετά τον πόλεμο του 2008 δεν έχει υπάρξει καμία διεθνή παρουσία στη Γεωργία. Η μόνη διεθνή παρουσία είναι η δική μας πολιτική αποστολή. Ούτε το Ρωμένα Έθνη, ούτε ο ΑΣΕ, ούτε το ΝΑΤΟ. Είμαστε η μόνη διεθνής παρουσία. Η αποστολή μας τι κάνει, να επιτηρεί τα διοικητικά σύνορα μεταξύ της Γεωργίας και των δύο αποσχιστήσεων περιοχών. Είναι οι μόνοι ανεξάρτητοι παρατηρητές επιτόπου. Και γιατί ήρθε χθε ο επικεφαλής, γιατί το τελευταίο δεκαπενθήμερο υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και φαίνεται ότι εν ώψη των εκλογών στη Γεωργία του χρόνου δυστυχώς θα επιδοθούν ακόμη περαιτέρω τα πράγματα. Έχουν ένα κόκκινο τηλέφωνο, αν υπάρξουν προβλήματα. Η αποστολή προσπαθεί να ηρεμήσει τους πάντες. Είναι σε επαφή και με τις δύο πλευρές. Έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και των δύο πλευρών. Και εγώ νομίζω ότι αν δεν ήσαν παρόντες, το ενδεχόμενο ένοπλης σύραξης, ακόμη και ατυχημάτων θα ήταν ε, πολύ υψηλότερο. Πολύ... Το ενδεχόμενο θα ήταν πολύ πιο πιθανό. Μπορώ να σας ε, περιγράψω ότι γίνεται σε κάθε αποστολή και λέω ότι κάθε μία είναι διαφορετική. Ορισμένες αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, όπως για παράδειγμα οι αποστολές μας στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να θέλουν και οι δύο πλευρές να συνομιλούν για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, απλώς τις ακυρώσαμε τις αποστολές και αποχωρήσαμε. Και κάθε έξι μήνες επανεξετάζονται. Το αποτέλεσμα της επανεξέτασης υποβάλλεται στα κράτη-μέλη και κάθε έξι μήνες τα κράτη-μέλη αποφασίζουν τι θα γίνει. Θα διατηρηθεί, θα συνεχιστεί ή αν δεν έχει πια έννοια γιατί ολοκλήρωσε την αποστολή της οι πλευρές δεν ενδιαφέρονται, οι εμπλεκόμενοι, τότε διακόπτεται η αποστολή αυτή. Είναι πάντα απόφαση των κρατομέλων. μελών. Τέλος. Ευχαριστώ για την ερώτηση που μου θέσατε. Η ερώτηση για τις επιπτώσεις ε, του Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα από τα 28 κράτη-μέλη. Έχει συμβάλει και στις στρατιωτικές και πολιτικές αποστολές μας. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει συμβάλει και τόσο πολύ. Δεν από τους πρώτους. Φυσικά θα έχει αρνητική επίπτωση και στις στρατιωτικές και τις άλλες. Η επίπτωση αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Εκεί που μπορεί να είναι πιο αξιοσημείωτη είναι στις στρατιωτικές αποστολές. Μία αποστολή, Αλτέα, στην Βοσνία Ζεγοβίνη είναι ε, μια αποστολή όπου το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα εφεδρικό τάγμα. Αν υπάρξει δραματική επιδείνωση της κατάστασης, το τάγμα αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για να στηρίξει την επιχείρηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διατεθειμένο να αφήσει αυτή την, αυτό το τάγμα εκεί, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Δεν μπορώ να σας πω τώρα πώς ακριβώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Αν είναι με συμφωνία η αποχώρηση, δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει διακανονισμός που να επιτρέψει να συνεχίσει να βοηθάει τον Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτή την αποστολή, αν είναι χωρίς συμφωνία. Θα ρωτήσουμε και έχουμε ήδη ρωτήσει τα κράτη-μέλη αν μπορούν να δώσουν περισσότερα. Αλλά όπως ξέρετε δεν είναι σαφής η κατάσταση σε αυτή τη φάση πώς και πότε θα υπάρξει αυτή η αποχώρηση. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε. Αλλά για τις πολιτικές αποστολές CSDP έχει συμβάλει πολύ λίγο το Ηνωμένο Βασιλείο, έχω εδώ τα στοιχεία. λιγότερο από 2%. Οπότε οι επιπτώσεις ε, δεν θα είναι και τόσο οδυνηρέ. Ευχαριστώ Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση αυτή, για την ειλικρίνεια και τη σαφήνεια με την οποία μας δώσετε τα στοιχεία αυτά είναι πολύτιμα για εμάς και θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε την ε, δουλειά μας, την συζήτησή μας σε αυτά τα ουσιαστικότατα στοιχεία σχετικά με τις αποστολές πολιτικής ασφαλείας της ε, κοινή πολιτικής. Ευχαριστούμε πολύ.